Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καθυστερήσαμε την έναρξη 15 λεπτά. Κλασικό για έναν Γερμανό θα έλεγε κανείς, αλλά ας ξεκινήσουμε την συνεδρίαση. Και αυτήν ξεκινήσουμε. πάρα πολύ σημαντικό έγγραφο που αφορά τον στόχο υπαριθμών 3. Μαρίτερε Σάντσε Σμίτ είναι η συγκίτρια. Πρόκειται για τον στόχο 3 που είναι πάρα πολύ σημαντική για την διασυνοριακή, διακρατική και περιφερειακή συνεργασία. Ο στόχο 3, η πρόκληση για δαφική συνεργασία. Και δίνω τον λόγο τώρα στην Μαρία Τερέ Σάντσε Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να δούμε το πρώτο slide λέει ο Μιλήτρια, που δεν βλέπουν οι διερμηνείς. Τώρα φαίνεται παντού η πρώτη διαφάνεια. Ωραία, τώρα μπορούμε να αρχίσουμε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η εδαφική συνεργασία είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ με ενδιαφέρει γιατί ζω σε μια διασυνοριακή χώρα, στο, πόλη στο Περπινιάν, της, κοντά στην Ισπανία. Και η συνεργασία για μένα επομένω είναι καθημερινή πρόκληση. Επίσης, το πρώτο εξάμεινο του 2006 συμμετέσχουν στη Γαλλία σε μια αποστολή που αφορούσε την διασυνοριακή συνεργασία ε, του κυρίου Φιλιών του Πρωθυπουργού. Η περιφέρεια μας επομένως ε, είναι εκτεθειμένη σε κάποιες ανισότητες, οπότε έχουν και τις δυσκολίες προσαρμογής της χώρας μας σε σχέση με την πρόκληση του ανοίγματο των συνόρων και της παγκοσμιοποίησης και της ολοκλήρωση. ολοκλήρωσης. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν φαίνονται διαφάνειες. Δεύτερη διαφάνεια. Ναι, εδώ αυτός ο χάρτη της χώρας και μπορείτε να δείτε τώρα τη μεταξύ των εργαζομένων και μπορείτε να δείτε την ε, ανισορροπία μεταξύ των δύο χωρών και σε αυτή την έκθεση προτείνουμε κάποια μέτρα για να βελτιωθεί η διασυνοριακή συνεργασία ούτως ώστε να φτάσουμε σε μια ισόρροπη ανάπτυξη για την περιφέρεια. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι δυνατόν ούτε το κράτος ούτε η περιφέρεια να αντιμετωπίσουν μόνοι του την, την πρόκληση αυτή. Χρειάζεται μια δυναμική ενεργειακή πολιτική και να σας πω ένα μικρό ιστορικό για να καταλάβετε τι ισχύει. Η Ευρώπη αποτελεί από 27 κρατημέλη και από 271 περιφέρειες και δυνάμει των διαφορετικών συνθήκων, όλο ένα και περισσότερα σύνορα έχουμε. Και με το Σέγγεν έχουν έρθει αυτά τα σύνορα, όμως ε, δεν έχουν έρθει τελείως γιατί στη καθημερινή ζωή το αντιμετωπίζουν οι πολίτες και με τα πολεμικά ε, έχουμε άτυπες συνεργασίες μεταξύ των περιφερειών. Αυτές οι συνεργασίες αντιστοιχούν στις διαφορετικές ανάγκες περιφερειών και πολιτών. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, προσπάθησε να απλουστεύσει τα πράγματα σχετικά με αυτό και έχουμε το Interreg και έτσι θεσμοθετήθηκε, ε, πλαισιώθηκε αυτή η συνεργασία. Πρόσφατα στο τουρνέ υπό την αιγύρια της Βελγικής Προεδρίας ε, γιορτάσαμε τα 20 χρόνια αυτής της συνεργασίας. Σε αυτά τα 20 χρόνια από ένα μικρό πρόγραμμα πρωτοβουλίας το Ιντερέγ έγινε ο στόχος 3 που αφορά την πολιτική συνοχή την περίοδο 2007-2013 και έχουμε ένα συγκεκριμένο νομικό εργαλείο που αφορά την ε, συνοχή των περιφερειών που τώρα είναι μια προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατοχυρώνεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας όπως η οικονομική και η κοινωνική συνοχή. Η συνεργασία επομένω τώρα αυτή έχει οριμάσει και γι' αυτό έχει αναπτυχθεί αυτή η προβληματική για τον στόχο 3 και θα ενταχθεί και στις ε, επόμενες συνομιλίες που αφορούν τον προϋπολογισμό. Ε, περιμένω τις προτάσεις σας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα αξιόλογο κείμενο με φιλοδοξίες που θα αντικατοπτρίζει την συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και έχουμε και αυτό το έγγραφο εργασίας, το οποίο είναι διερευνητικό περισσότερο για να πείτε τη γνώμη σας και να καταλήξουμε σε κάποια ξεκάθαρη στάση του Κοινοβουλίου με συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον του στόχου 3. Τρίτη διαφάνεια. Το πρώτο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να τεθεί είναι το εξής. Ποιες είναι οι στρατηγικές φιλοδοξίες που θα πρέπει να καλυφθούν από την διαπεριφερειακή συνεργασία. Αν δεν έχουμε σαφείς στόχους δεν γίνεται τίποτα και για μένα η διαπεριφερειακή συνεργασία θα πρέπει να άρει τα σύνορα και θα πρέπει να οικοδομήσει την Ευρώπη με την καθημερινή ζωή. Να μην έχουμε μόνο φραγμούς και έτσι όλοι μαζί, περιφέρειες ε, και, κράτη, να προχωρήσουν και έχουμε κάποιους επικρίσεις κατά του στόχου 3, το ότι δεν υπάρχει εμβέλεια στατικική και δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση, οπότε ε, θεωρούν ότι η συνεργασία αυτή είναι κάπως φλού, αόριστη και δεν υπάρχουν κάποια μετρήσιμοι στόχοι. Επίσης θα χρειάζεται να υπάρχει ένα στρατηγικό πλαίσιο σημαντικό και όλοι να μπορούν να συμμετάσχουν με όλες τις πολιτικές της Ευρώπης και με την στρατηγική ενώπιση του 2020 θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στην περιφερειακή συνεργασία της οποίας ο ρόλος θα είναι να συνεργαστούν οι περιφέρειες σε σχέση με την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων, ε, ψηφιακή τεχνολογία, περιβάλλον, μεταφορές. Παρ' όλα αυτά ε, έχουμε περικοπή των, ε, των πόρων και η μικρή αυτή προοικοδότηση θα πρέπει να φρενάρει μια τέτοια σημαντική εξέλιξη. Επομένως χρειάζεται μια, μια στατική bottom-up να εμπλακούν οι τοπικοί παράγοντες γιατί υπάρχει άνηση ε, ε πρόοδος. Το Βέλγιο και η Γαλλία έχουν μια τέτοια παράδοση συνεργασίας, αλλά αυτό δεν ισχύει παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχουν κάποιοι, κάποια όρια ε, ανάλογα με την περιφέρεια. Ε, άλλα στη Σιλεσία, στην Πολωνία, άλλα στο Πούι, στην ε, Ιταλία. Άρα χρειάζονται πλέον κάποια κίνητρα οικονομικά για αυτούς οι οποίοι εμπλέγονται, ούτως ώστε με συγκεκριμένο τρόπο να καλύπτουν, καλύπτουν τα κριτήρια για τους στόχους Ευρώπης 2020. Άρα αν αυτά τα 7,5 δις για τον στόχο 3 και για την περίοδο 2007-2013 είναι κάτι το σημαντικό είναι παρόλα αυτά μόνο το 2,5% της πολιτικής συνοχής. Ε, στόχος 1 είναι 250 δις και ε, την άλλη εδώ είναι πολύ λιγότερα αυτά που ζητούμε και ο στόχος 3 καλύπτει όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι δίνονται δυνατότητες προσέγγισης ούτω ώστε είναι δυνατόν χώρες και πολίτες να βοηθήσουν και να έχουμε μια προσθεμένη αξία διότι ο στόχος 3 ε, συμβάλλει ε, στην πιο στενή ε, ένωση προσέγγιση των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να δούμε και το επόμενο ερωτήμα που αναδιώνεται. Ποια θα πρέπει να είναι η δημοσιονομική κατάσταση όσον αφορά το στόχο 3 και τους άλλους δύο στόχους. Ε, ξέρω ότι τώρα εξελίσσεται ζήτηση δημοσιονομικά και ακόμα δεν έχουμε καθορίσει τα σχετικά ποσά. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένας, ε, ε, ένα ποσό και δεν θα πρέπει να, να είναι όμοιρος αυτός ο στόχος σε σχέση με άλλα κονδύλια. Θα πρέπει επομένω να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε αυτή την προσθέμενη αξία, τι να κάνουμε όσον αφορά το πώς αυτά που ε, ξοδεύουμε σε νοσιακό επίπεδο θα αποδίδουν περισσότερα από σε εθνικό επίπεδο. Εδώ υπάρχει μεγάλη προσθέμενη αξία και θα πρέπει να δούμε με ποιον πιο αποτελεσματικό τρόπο θα φτάσουμε σε μια ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Να γίνει όσο γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων. Θα πρέπει να δούμε πώς θα συνδυαστεί ο στόχος 3 με τους άλλους δύο στόχους. Συνέργεια, ούτως ώστε να κάποια λειτουργικά προγράμματα για πολλές περιφέρειες διασυνοριακά θα τα χρησιμοποιήσουμε, τα οποία να ε, αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα θέματα, θεματικά κεφάλαια όπως τη Γαλλία και άρα θα πρέπει τώρα να αναθεωρήσουμε κάποιες διατάξεις του ΦΕΝΤΕΡ. Τέλος, όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να ενθαρρύνουμε μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ διαφορετικών στόχων, συνεργασία διασυνοριακή, διαπεριφερειακή και κάποια μέσα όπως ένα ευρωπαϊκό μέσο πολιτικής γυτνίασης ή για την προενταξιακή φάση. Η αρχιτεκτονική του, του στόχου 3 είναι ως εξής τώρα, διασυνοριακό 73%, ε, διακρατικό 20% και διαπεριφερειακό που είναι 4% των πιστώσεων και τρία προγράμματα Urbact, Interact και Spon. Για δούμε, αυτή η αρχιτεκτονική θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει έκτη διαφάνεια. Και τώρα μπορείτε να δείτε τι ισχύει όσον αφορά την διασυνοριακή συνεργασία. Από πλευρά μου, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να μείνει αυτή η διάκριση με διαφορετικών πτυχών τη συνεργασία με κάποιε διευθετήσει και αν χρειάζεται να γίνει κάποια αλλαγή, θα πρέπει να προσέξουμε να μην τεθούν ένα αμφιβόλο τα όσα έχουν μέχρι σήμερα επιτευχθεί. Επίση θα πρέπει έτσι να δούμε πώς θα έχουμε καλύτερο συντονισμό και διακυβέρνηση όπως ταιριάζει για τις στρατηγικές μας. Έβδομη διαφάνεια. Να εδώ ένα παράδειγμα της ε, διακρατικής συνεργασίας, θα πρέπει να γίνει καλή συντονισμό της μακροπεριφερειακής συνεργασίας σε σχέση με τον στόχο 3 του διακρατικό και αυτό θα πρέπει να εξελιχθεί. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η μακροπεριφέρεια είναι μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου και εδώ η λογική είναι λογική συντονισμού, ένα σχέδιο κοινό που το οποίο αφορά πάρα πολύ μεγάλα εδάφη και έτσι έχουμε εδώ κάποια πλεονεκτήματα ολοκληρωμένης πολυκλαδικής προσέγγιση με μια στρατηγική δράση επί τη βάση υπαρχόντων πόρων. Να μην ισχύει το κριτήριο των 150 χιλιόμετρων όσον αφορά τι απομακρυσμένε νήσους και ε, επικράτειες. Ε, ε, αυτό το έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο στο σχετικό ψήφισμα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, των αεροκατημένων περιοχών. Οπότε, τέλος, έχουμε μια μελέτη που ζήτησε να γίνει το Κοινοβούλιο όσον αφορά αν μπορεί να έχουμε κάτι σαν έρασμος για τους ερετούς άρχοντες και να δούμε πώς μπορεί το Interreg να βοηθήσει τις σχετικές ανταλλαγές, το URBAC και η διακρατική συνεργασία βοηθούν στο να υπάρξει ένα δίκτυο τέτοιο που να βοηθά στο μέλλον το φιλόδοξο αυτό ε, πρόγραμμα, αυτή την εκδοχή του έρασμου. Ο στόχος 3 έχει κάποια νέα νομοθετήματα, νομοθετικά εργαλεία για να διευκολύνει την υλοποίηση αυτού του είδους την ομαδοποίηση της διπεριφερειακής συνεργασίας. Και να ένα παράδειγμα από τη χώρα μου και έτσι είναι δυνατόν οι τοπικοί, περιφερειακοί σε διάφορα επίπεδα να ομαδοποιούνται, να έχουν νομική προσωπικότητα και να μπορούν να φέρουν πέρα κάποια προγράμματα και αυτές είναι οι ανάγκες που θα πρέπει να αντιστοιχούν στο νομικό πλαίσιο, στην δημοσιονομική προοικοδότηση. με αυτά τα συμβούλια, τα διακρατικά και διαπεριφερειακά. Και έτσι η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και να καλύπτει αυτές τις ομαδοποίησεις. Ένατη διαφάνεια. Μετά από αυτή την, την πορεία θα πρέπει να δούμε τι διαχείριση έχει γίνει όσον αφορά τις συμβάσεις τις αναπτυξιακές για τους στόχους εν του 2020. Είναι πολύπλοκη η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων και πολλές φορές ε, εμφανίζεται, άρα θα πρέπει να απλουστευτεί η διαδικασία και να μην αποθαρρύνουμε αυτούς που ασχολούνται με τα προγράμματα. Επόμενη διαφάνεια. Θα πρέπει να μην έχουν τι αντιδράσει του τύπου θέλω πίσω τα λεφτά μου. Και ο καθένα επομένω ανακαλεί κάποια την, την εισφορά του και ενεργεί μόνος του. Χρειάζονται επομένω έλεγχοι, οικονομική έλεγχη από την κάθε πλευρά. Θα πρέπει να δούμε πώς το κόστος θα κατανεμηθεί με πιο απλό τρόπο θα πρέπει να έχουμε κάποιες προθεσμίες κατάλληλες για να διευκολύνουν τους διαχειριζόμενους τα κονδύλια. Το Ευρωβαρόμετρο ε, έδειξε ότι 80% των Ευρωπαίων ποτέ δεν άκουσαν για την διαπεριφερειακή συνεργασία. Θα πρέπει για τους χρήστες όλα αυτά να είναι φιλικά, θα πρέπει να, είναι, να έχει προβληθεί πιο ορατό αυτό το αυτή η υπόθεση και να γίνει ανάλογος προγραμματισμός και εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών σε κάθε επίπεδο. Και έτσι αυτές οι πολιτικές να έχουν προβληθεί περισσότερο ως προς τον κόσμο. Ενδέκατη διαφάνεια. Θέλω τις ε, ιδέες σας, ούτως ώστε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον με τον στόχο 3. Η επόμενη διαφάνεια, σας ευχαριστώ. Αλλά πάμε πίσω τώρα στο 11. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Κυρία Σάντσες Σμιτ. Υποστηρίζεται με θέρμη και ενθουσιασμό την διαμεθοριακή συνεργασία για όλους μας εδώ, όλες και όλους, Χρειάζεται ακόμα συζήτηση των διαφόρων στόχων. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαϊτέ Σάντζε Σμιτ για την ποιότητα τη δουλειά τη σε σχέση με τον στόχο 3 και το μέλλον και με χαρά την άκουσα να μιλά για τη συμμετοχή των ε, τοπικών ε, φορέων, των τοπικών αρχών. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την αξιοποίηση της πολιτικής συνοχής στις διάφορες περιφέρειες και με τους πολίτες, με την ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα στους διάφορους τοπικούς ε, άρχοντες ε, των κρατών μελών. Έχω δουλέψει λοιπόν με το έρασμος των ε, τοπικών αρχών και των τομικών αρχόντων και ακριβώς στο πλαίσιο ενός προγράμματος πιλότου, γιατί έχουμε μια πρόβλεψη 2 εκατομμυρίων ευρώ για να ξεκινήσει ένα πρώτο πρόγραμμα που θα ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Και έχω προτείνει διάφορους σε διάφορους ε, εμπλεκόμενους αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δουλέψουμε πάνω σε ένα πλωτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο των διαμεθοριακών ή ε, διακρατικών σχέσεων. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν πολύ μια κοινή ε, συνεργασία για να δούμε από κοινού πώς θα μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή αυτό το έρασμος των τοπικών αρχόντων μέσω του Interreg. Και το δεύτερο που θα ήθελα επίσης να δούμε είναι η πτυχή πολίτης αυτού του εγχειρήματο που νομίζω ότι είναι ε, σημαντικό. Νομίζω πως ε, πολλές φορές μένουμε πολύ σε τεχνοκρατικά και νομικά ζητήματα ε, και οι πολίτες δεν εμπλέκονται. Είναι εργαλεία τα οποία δεν τα γνωρίζουν αρκετά οι πολίτες και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτές οι δομές οι οποίες αξιοποιούν τα διάφορα προγράμματα του στόχου 3 αυτές τις δομές να τις ιδιοποιηθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες, να γνωρίζουν πόσο παρούσα είναι η Ευρώπη στις ε, περιφέρειες, πόσο συμμετέχει στη δημιουργία απασχόλησης, επιχειρήσεων, στην ε, διαχείριση των δομών, ώστε να βελτιώσει την καθημερινή του ζωή, αλλά και το μέλλον τους. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καντέκ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με την ευκαιρία της παρουσιάσεως θα τονίσω τη σημασία της διαπεριφερειακής στρατηγικής. Ευχαριστώ βέβαια και τον εισηγητή για το έγγραφο εργασία που θέτει το θέμα του συντονισμού μεταξύ του στόχου 3 και των στρατηγικών διαπεριφερειακής συνεργασίας. Ο στόχος 3 είναι παρκές πλαίσιο. Πρέπει να στραφεί γύρω από στόχους κοινούς με κοινά χαρακτηριστικά και γεωγραφικά στοιχεία. Σήμερα η περιφέρεια της Βαλτικής προχωρεί σε μια μακροπεριφερειακή συνεργασία, αργότερα η περιοχή του Δούναβη. Οι μακροπεριφέρειες είναι εύκαμπτο πλαίσιο συνεργασίας, χωρίς έξτρα επιβάρυνση για τις ε, κοινότητες, δεν δημιουργεί νέους θεσμούς, ούτε νέα νομοθεσία. Επομένως εντάσσεται στα πλαίσια του στόχου 3. Το ερώτημα είναι, χρειάζεται, αν παραμείνει ο προπολογισμό όσο έχει, να φτιαχτεί ειδικό κονδύλιο στην επόμενη δημοσιονομική προοπτική ή μάλλον πρέπει να συνδυαστούν, ή να συνδεθούν μάλλον οι στρατηγικές αυτές μακροπεριφερειακές με τον στόχο 3. Η διάσταση αυτή προσφέρει μια προστιθέμενη αξία. Επίσης οι μακροπεριφερειακές συνεργασίες πρέπει να βασιστούν σε αποτελεσματικές διαρθρώσεις ανάμεσα στις εθνικές αρχές και στις τοπικές αρχές με συνεργασία βέβαια των ευρωπαϊκών αρχών. Όπως εξήγησαν προηγουμένως οι συνάδελφοί μου, η σωστή διαχείριση μπορεί και να εφαρμοστεί και στη μακροπεριφερειακή συνεργασία. Χρειάζεται ένα απλό πλαίσιο για μια αποδοτική μακροπεριφερική συνεργασία. Άρα, μας ενδιαφέρει να δώσουμε μέσα στο στόχο 3 μια ε, εντονότερη διάσταση των ε, μακροπεριφερειακών συνεργασιών για να επιτύχουμε τους στόχους που προανέφερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κατέκ. Ο κύριος Κέλλη. Συγχαρητήρια και από τη δική μου πλευρά για την κυρία Σάντσε Σμιθ. Σπουδαία γυναίκα λέμε εμεί στην Ιρλανδία για κάτι τέτοιε. Νομίζω ότι χρειάζεται και άλλη συζήτηση και θα έχουμε την ευκαιρία να το πράξουμε. Είπε ότι μόνο 2,5% του Ταμείου Συνοχής πηγαίνει στον στόχο 3. Και είπε ότι πρέπει να εξεταστεί η διασύνδεση μεταξύ των τριών στόχων ώστε να ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό, μίλησε η κυρία Σάντζε Σμιθ, για την διάθεση κονδυλίων με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται εσωτερικές διαμάχες και να δίνεται ένας ε, εντονότερος ευρωπαϊκός χαρακτήρας με εξοικονόμηση και κόστους. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να εγκύψουμε σε αυτά για να τα συζητήσουμε κι άλλο και να λάβουμε και άλλες αποφάσεις ώστε να εξασφαλίσουμε προστιθέμενη αξία ε, σε οποιοδήποτε δαπάνες εγκρίνουμε για στόχους 3. Άρα υπάρχει ανάγκη περαιτέρω συζητήσεων βασισμένο σε, αυτή, σε αυτές τις σωστές συστάσεις. Μπράβο και πάλι. Πρόεδρο σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προέρχομαι και αξίζει να το πω από μια περιοχή του Ρήνου που είναι η παλαιότερη ευρωπεριφέρεια στα βέλγο-γερμανικά σύνορα με εξαιρετικές εμπειρίες από τη συνεργασία αυτή. Εγώ θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο αυτό που είπε ο κ. Καντέκ, η επέκταση δηλαδή στις μακροπεριφέρειες. Διότι προκαλούνται δυσχέρειες από τις αυξημένες αξιώσεις που έχουν οι περιφέρειες αυτές και είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις παραμεθόριες περιοχές να διατίθεται κονδύλια του Interreg. Ναι, μεν τα σύνορα δεν υπάρχουν πλέον στα χαρτιά, αλλά σε πολλά καθημερινά θέματα τα οποία αφορούν τη μετακίνηση από τη μία πλευρά των συνόρων στην άλλη. Εξακολουθούν να σημειώνονται προβλήματα, ακόμα δεν έχουν επιληθεί. Χρειάζεται λοιπόν, χρειάζονται λοιπόν μηχανισμοί οι οποίοι να λειτουργούν σωστά. Χρειάζεται να εγκύψουμε σε αυτά, αυτό είναι σαφές, αλλά αυτό η προσπάθεια δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρος του προβληματισμού που εξακολουθούμε να έχουμε και των προβλημάτων που εξακολουθούμε να έχουμε σε παραμυθόριες περιοχές. Ευχαριστώ. Διαφαίνεται μια ακόμα ενδεχόμενη σύγκρουση. Μέχρι τώρα ζήτησαν το λόγο μόνο συνάδελφοι του Λαϊκού Κόμματος. Χαίρομαι τώρα που ζητεί το λόγο ο κ. Βλάζακ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ με τη σειρά μου την εισηγήτρια για το έργο της και για την παρουσίασή της, στην οποία παρουσίαση έθιξε ορισμένα σημαντικά θέματα και εγώ θα έλθω σε δύο από αυτά. Πρώτον, την αύξηση της γνώσης και της συνείδησης για τη σημασία τη διαμεθορικής συνεργασία καθώς και την αύξηση της γνώσης για το πώς μπορούν να επιτύχουν οι ενδιαφερόμενοι χρηματοδότηση. Αυτό βέβαια είναι σημαντικό ιδίω για του τοπικούς άρχοντες. Είναι κάτι το οποίο για πολύ καιρό επιδιώκει άλλωστε η Επιτροπή μας. Το δεύτερο που θέλω να θέσω είναι οι συζητήσεις μεταξύ τοπικών εκπροσώπων, περιφερειακών εκπροσώπων εθνικών ε, αρχών ή εθνικών πολιτικών ανδρών και ευρωπαϊκών. Πρέπει να γνωρίζουμε αν υπάρχουν διαφορές επιτόπου στην περιφέρεια. Να μπορούμε να συγκρίνουμε τις απόψεις με ταξί των διαφόρων επιπέδων τοπικού, περιφερειακού και ευρωπαϊκού, εθνικού μάλλον και ευρωπαϊκού. Σας ευχαριστώ για την ε, πρόταση αυτή. Ο κύριος Αλφόνση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να εκφράσω το ενδιαφέρον της ομάδας μας για την έκθεση αυτή. Όντως τα σύνορα και η διασυνοριακή συνεργασία είναι αναμφισβήτητα το, ο χώρος όπου είναι πιο προφανή τα κοιτάσματα παραγωγικότητας για την Ευρώπη. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση για αυτό το νοσοκομείο που επιτρέπει στους βόρειους και στους νότιους Καταλανούς να μοιράζονται ένα νοσοκομείο ενώ ήταν όλοι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν πολύ πιο μακριά. Ένα επιτυχημένο λοιπόν παράδειγμα. Πόσα όμως ε, αντίθετα παραδείγματα ξέρουμε, ξέρουμε ας πούμε γιατί η χώρα των Βάσκων υπάρχει ένα μεγάλο ε, ε, αεροδρόμιο στο Μπιαρίτς και από την άλλη πλευρά στην Ισπανία έχουμε άλλο ένα μεγάλο αεροδρόμιο αν κάνουμε το γύρο της Ευρώπης θα δούμε πολλά τέτοια παραδείγματα και γι' αυτό ακριβώς και είναι σημαντικό να ασχοληθούμε καθώς μάλιστα τα κράτη-μέλη έχουν, έχουν οικοδομηθεί γύρω από αυτά τα σύνορα και δεν έχουν πάντοτε τα απαραίτητα τα για να προχωρήσουν και ακριβώς αυτό είναι η ευρωπαϊκή επικουρικότητα που θα πρέπει να εφαρμοστεί. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε το μήνυμα και να προωθήσουμε αυτό το ε, ντοσιέ. Όσον αφορά τώρα συγκεκριμένες προτάσεις, νομίζω θα πρέπει να ασχοληθούμε για να διευκρινίσουμε τις δυνατότητες τις ευρωπεριφέρειες, μακροπεριφέρειες και τα μεγάλα προγράμματα περί προβληματισμού και συντονισμού, τα πραγματικά λειτουργικά εργαλεία που επιτρέπουν να γίνει συνεργασία ανάμεσα στους θεσμούς, είτε πολύ συγκεκριμένα προγράμματα, ένα νοσοκομείο, η προστασία της ε, βιοποικιλότητα. Δεν έχουμε ίσω αποσαφηνίσει πολύ ε, διάφορα εργαλεία, πάντως θα πρέπει να ασχοληθούμε με τη λειτουργικότητα καθενό από αυτά τα εργαλεία και, να κάνουμε και θα κάνουμε και συγκεκριμένε τροπολογίες προ αυτή την κατεύθυνση. Σα ευχαριστώ κύριε Αλφονσί, σκιώδης ηγητής των Πρασίνων, ο κύριος Μάτουλα. Ευχαριστώ. Συγχαίρω την συνάδελφό μας κυρία Σάντσε Σμιτ για την ιδέα που είχε, για την επιλογή του πολύ ενδιαφέροντος θέματος και να μου επιτρέψει να προσθέσω λίγες σκέψεις μου σχετικά με την Ανατολική Ευρώπη και κυρίως τα σύνορα μεταξύ Ρουμανίας και Ουγγαρίας που ε, είναι η περιφέρεια από την οποία προέρχομαι και που νομίζω ότι ωστόσο αφορούν και άλλες περιφέρειες. Η υποστήριξη ενός προγράμματος έρασμος για τους τοπικούς άρχοντες. Ναι, γιατί. Διότι τα τελευταία 20 χρόνια στην Ανατολική Ευρώπη εμείς έχουμε επιτελέσει θαύματα. Μην λησμονούμε ότι ακόμα πριν από 20 χρόνια υπήρχε το σιδηρούν τείχος και προέκυψαν σημαντικότατες αλλαγές μετά την πτώση του. Νομίζω ότι οι τοπικοί άρχοντες, οι τοπικοί εκλεγμένοι άρχοντες στην διαμεθορική συνεργασία έχουν λάβει αποφάσεις που έχουν φτάσει μέχρι και να επηρεάσουν τις εθνικές πολιτικές αποφάσεις. Στην αρχή είχαμε πολύ λίγα κονδύλια στη διάθεσή μας. Αλλά αυξάνει σιγά σιγά ο όγκος τους. Η μεγάλη πλειοψηφία των πρωτοβουλειών που γνωρίζω έχουν τοπικό χαρακτήρα. Στην περιφέρειά μου υπήρξε, για παράδειγμα, μια συνεργασία μεταξύ των αρχών ανάμεσα στα, μάλλον εκατέρωθεν των συνόρων, για την υδροδότηση με πόσιμο ε, νερό. Από τη μια χώρα στην άλλη. Το ίδιο ισχύει για την κινητικότητα των εργαζόμενων στις ε, παραμεθόριες περιοχές. Η κινητικότητα αυτή έχει αυξηθεί σημαντικά. Προ 15 ετών δεν θα μπορούσαμε καν να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Σήμερα όχι μόνο υπάρχει, αλλά όπως είπα αυξάνεται. Γνωρίζουμε βέβαια ότι είναι δύσκολο να τροποποιηθεί η δομή του προπολογισμού. Ωστόσο υποστηρίζω την ιδέα που λέει ότι χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια διότι τα χρήματα αυτά πιάνουν τόπο εν τέλει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Σίμων. Θα συμφωνήσω με την κυρία Φερχάιν. Εάν ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτό των μακροπεριφερειών όπως της Βαλτικής ή του Δούναβη που ε, βρέχει και τη δική μου περιφέρεια, δηλαδή να δώσουμε ιδιαίτερα κονδύλια από τον προπολογισμό, τότε δίνουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα στι περιφέρειε αυτέ. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε από τον στόχο 2 ε, προγράμματα ε, κατά μήκο του Δούναβη ή στην ε, περιφέρεια της Βαλτικής. Μετά μπορούμε να ενισχύσουμε, για παράδειγμα, διασκέψεις, διοικητικέ προσπάθειες. Αυτό είναι σκόπιμο. Μπορούμε να φροντίσουμε αλλά αυτά τα ε, προγράμματα πρέπει να μπορούν να υποβάλουν σε αιτήσει χρηματοδότηση μέσα στα πλαίσια του προγράμματος 3, αλλά να τους δοθεί έξτρα βαρύτητα απέναντι σε άλλες περιφέρειες δεν θεωρώ ότι είναι σκόπιμο, ούτε ενδεδειγμένο, διότι υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες συνεργασίας οι οποίες φτάνουν στο ύψος και της ε, συνεργασίας των Δουναβία. Πρόεδρος, Κανείς άλλος. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κανείς άλλος που επιθυμεί να λάβει το λόγο. Ας δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος επιθυμεί να τον λάβει για το θέμα αυτό. Όχι. Καλά λοιπόν. Τότε θα δώσω τον λόγο πάλι στον συντονιστή του Λαϊκού Κόμματος και μετά να ολοκληρώσει η συγγύτρια. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι. Διάβασα το έγγραφο με μεγάλο ενδιαφέρον. Εάν υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή προστιθέμενη τότε είμαι βέβαιος ότι αυτή βρίσκεται στην ε, διαμεθοριακή συνεργασία. Όπου και από τις δύο πλευρές των συνόρων μπορούν να επιτευχθούν πολλά σημαντικά πράγματα που έτσι προσθέτουν αξία. Αυτή η συνεργασία λοιπόν, όπως είπα, προσφέρει σημαντική αξία. Ωστόσο, θα ήθελα να προσθέσω, να κάνω ένα βήμα παραπέρα και να θέσω υπόψη σας την εξής σκέψη. Συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, δηλαδή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. Θέμα το οποίο πρόσφατα θέσαμε ως ερώτηση στην Ολομέλεια και μας απάντησαν ότι τέλη του τρέχοντος έτους, αρχές του επομένου έτους θα έχουμε κάποιες πρώτες αξιολογήσεις για τη συνεργασία αυτή. Υπάρχουν ακόμα σημαντικά ερωτηματικά σε ό,τι αφορά τον τρόπο πρόθεσης, την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Ωστόσο, πρέπει να συγκρίνουμε την οικονομική επιβάρηση που θα προκύψει με το όφελος που προκύπτει από τη διαμεθορική συνεργασία. Επίσης, το μοντέλο συνεργασίας που έχουμε μέσα στην ίδια την Ευρώπη μπορεί να διευρυνθεί έτσι ώστε να περιλάβει και περιφέρειες οι οποίες δεν είναι ακριβώς στη Μεθόριο. Αλλά Στο στόχο 3 θα μπορούσε να γίνει, στα πλαίσια του στόχου 3 θα μπορούσε να γίνει αυτή η συζήτηση και ένα μέρος του προϋπολογισμού να ε, διατεθεί στην ε, προσπάθεια αυτή. Επισκέφθηκα την Κίνα πριν από λίγες ημέρες και <clears throat> είδα ότι το μέγα πρόβλημα εκεί έγκυται το ότι σε ορισμένες περιφέρειες της χώρας αυτής αυξάνει σημαντικά η κοινωνική ευημερία, ενώ αλλού όχι. Και δεν υπάρχει τρόπος να εξισορροπηθεί, δηλαδή να μεταφερθεί από τη μία περιφέρεια σε άλλη. Ευχαριστώ. Τελικά η κυρία Σάντσε Σμιτ θα λάβει ξανά το λόγο, η συγγετρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι αρκετά ικανοποιημένη και ευτυχής που βλέπω ότι Όποια και αν είναι η χώρα προέλευση η πολιτική ομάδα των ε, συναδέλφων, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ε, για την προστιθέμενη αξία αυτής ε, της πολιτικής. Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο να δείξουμε πως η πολιτική συνεργασία είναι ένας τρόπος να εφαρμόσουμε την Ευρώπη με συγκεκριμένο τρόπο. Να απαντήσω και στον κύριο Αλφόνση. Νομίζω ότι στο πλαίσιο της ε, δαφικής συνεργασίας δεν έχουμε επιλέξει πολύ μεγάλα προγράμματα ή εργαλεία ή συγκεκριμένα εργαλεία. Μάλλον θα πρέπει να βρούμε ένα μείγμα, ένα κατάλληλο μείγμα ανάμεσα στις διάφορες προτάσεις που υπάρχουν σήμερα γιατί οι περιφέρειες διαφέρουν, οι πρακτικές είναι διαφορετικές επίσης. Η γεωγραφική κατάσταση της κάθε περιοχής επίσης διαφέρει. Θα πρέπει να βρούμε δηλαδή τα κατάλληλα και προσαρμόσιμα εργαλεία. Ε, διαπίστωσα επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για το έρασμος των ε, τοπικών αρχών. Ε, θα πρέπει αυτό να το βάλουμε ε, σε εφαρμογή, να μπορέσουν να ανταλλάξουν τις πρακτικές τους, να μπορέσουν οι τοπικές μας αρχές και οι πολίτες μας να ιδιοποιηθούν ίσως αυτή την πολιτικοί εκμεταλλευόμενοι τις εμπειρίες που έχουν ήδη γίνει. Ε, επίσης σημείωσα το, η πρόταση της κυρίας Ανκών να κάνουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Την ανάγκη για περισσότερα χρήματα. Δυστυχώς δεν νομίζω πως είναι ευνοϊκή η κατάσταση θα πρέπει να επιμείνουμε στο να διατηρηθεί ίσω και να αυξηθεί ο προπολογισμό. Νομίζω πω θα γίνει μια συζήτηση για την ισορροπία των στόχων κυρίως με ένα στόχο σύγκληση, γιατί ε, ξέρουμε ότι θα αλλάξει η κατάσταση και από ό,τι κατάλαβα το θέμα των μακροπεριφερειών είναι επίσης σημαντικό. Θα πρέπει και σε αυτό να κρατήσουμε μια ξεκάθαρη θέση. Δηλαδή να δούμε αν είναι απαραίτητο να γενικευθεί ή να αφήσουμε τις ε, πρωτοβουλίες ε, στις περιφέρειες. Να, να ομαδοποιηθούν σε μακροπεριφέρειες, αν αισθανθούν αυτή την ανάγκη. Αν το καθιστούν απαραίτητο δηλαδή τα κριτήρια ή τα προγράμματα. Αλλά δεν νομίζω πως πρέπει να γίνει γενικευμένα αυτό σε όλη την επικράτεια. Αυτά είναι τα στοιχεία πάντως που εγώ κατέγραψα και που θα προσπαθήσω να τονίσω στην έκθεσή μου. Τώρα προφανώς ε, είμαι υπέρ, αλλά ε, μάλλον και δέχομαι τις δικές σας προτάσεις, τη συμβολή σας ε, για αυτή την έκθεση για το στόχο 3. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Okay, thank you very much, Σας ευχαριστώ κυρία Σάντσε Σμιτ. Η συζήτηση αυτή θα πρέπει τώρα να ολοκληρωθεί εδώ και νομίζω σε λίγα λεπτά θα αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ. Dear colleagues, we will be... αρχίσουμε την ψηφοφορία σε ένα λεπτό. Αυτό το λεφτά μια το εδώ το χρησιμοποιήσω για να σα ενημερώσω όσον αφορά τι αποφάσει που ελήφθησαν χθε από του συντονιστάς. Και σα ενημερώνω τι θα γίνει όσον αφορά το ποιο θα αναλάβει ποια γνωμοδότηση. Έχουμε γνωμοδότηση για το σχέδιο οργανισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για συγκεκριμένα μέτρα της Γεωργίας στις, στην απότερη περιφέρεια της Ένωσης. Αυτό το πήρε η Γκουε κατόπιν την ενίσχυση της ε, ανάπτυξης της υπαίθρου και το σχετικό ταμείο. Αυτό το ανέλαβε το ΕΛΚ. Ευρωπαϊκή Ευρωζωνικότητα επίσης το ΕΛΚ. Κινητοποίηση του Ταμείου αλληλεγγύης για Ιρλανδία, Πορτογαλία, Μαδέρα και Γαλλία αποφασίστηκε λόγω πίεσης χρόνου ότι η πρόεδρό σας θα στείλει επιστολή και όποιος ε, ενδιαφέρεται να διαμορφώσει την επιστολή μπορεί να μας πει τη γνώμη του και όσον αφορά την καινοτομία στην Ένωση αποφασίστηκε ε, η πρόεδρος να την κάνει και μη νομοθετικές εκθέσεις στα πλαίσια επίσης της ε, μελλοντικής μας πολιτικής αποφασίστηκε το ΕΛΚ να το αναλάβει όσον αφορά την ε, πολιτική συνοχή για το μέλλον επίσης αποφάσισαν οι συντονιστές οι πράσινοι να προτείνουν ένα θέμα για, προ... για έκθεση δίας πρωτοβουλίας αρχές 2011 και στη συνέχεια η γραμματεία πρόκειται να ενημερώσει τους συντονιστές όσο γίνεται συντομότερα όσον αφορά τις ανακοινώσεις Επιτροπής. Το ίδιο και όσον αφορά το σχέδιο κανονισμών για το επόμενο νομοθετικό πακέτο και έτσι θα ενημερωθούν όλοι από τη γραμματεία. Επίσης αποφασίστηκε τώρα η ομάδα να μελετήσει το τι μελέτες θα γίνουν το 2011 και επίσης είπαμε να χρησιμοποιήσουμε την συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα για εμπειρογνωμοσύνες που χρειάζονται και επίσης αποφασίσαμε να Α, όχι, συγγνώμη. Είπαμε να γίνει μια έκτακτη συνεδρίαση στα πράγματα, στα πλαίσια της έκθεσης της Πέμπτης για την Συνοχή. Και θα σε επαφή με την Επιτροπή όταν εγκριθεί αυτό το κείμενο. Δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα, αλλά είπαμε να γίνει μια τέτοια έκτακτη συνεδρίαση αρχάς Νοεμβρίου. Επίσης, να αναβληθεί ψήφιση για το σημείο 9 της Μερσίας Διατάξεως και να γίνει η ψηφοφορία στην έκτακτη συνεδρίαση. Είπαμε ότι συμφωνούμε στα όσα κατέληξε η ομάδα εργασίας. Να ετοιμαστεί ένα έγγραφο για την παρέμβαση της Προέδρου στο Φόρουμ Συνοχής των Βρυξελών στις 31 πρώτου και πρώτη Δευτέρου. Αυτές είναι οι προτάσεις των συντονιστών και ελπίζω ότι τις εγκρίνεται. Μπορούμε τώρα να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Δεν θα είναι εύκολη, αλλά πρέπει να γίνει ο έλεγχος πρώτα-πρώτα το αν λειτουργούν οι συσκευές και οι κάρτες ψηφοφορίας, να κάνουμε μια δοκιμή, ψηφίζουμε, ψηφίστε. The... Can we close? close. Πέρασε. Εψήφισαν όλοι, όλοι εντάξει. We can start uh, our vote. The first vote is on uh, Petru Konstantin Luhan. Uh, η πρώτη έκθεση. Πέτρο Κωνσταντιν Λούχαν για την επίτευξη εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, απαραίτητη προπόθεση για την ανταγωνιστικότητα. Αυτό με ερωτηματικό. Το ερωτηματικό θα παραμείνει, το έχω εδώ στο τέλος του τίτλου της έκθεσης και να αρχίσουμε ψηφορία. 15 συμβαστικές. Τρίτη, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 4. Πίνει υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος. Και τώρα θα γίνει έλεγχος στην 31. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 25-18. 34. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 46 καταπίπτει. Συμβαστική 9. Ε, ναι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κύριε Ματσόνη. Πρόεδρε, συγγνώμη, για τη σύνδεση της τροπολογίας 46 με τη συμβαστική 4 και τη συμβαστική 7, εγώ έχω απορίες, γιατί επί της ουσίας δεν υπάρχει καμιά αντίθεση. Γιατί λοιπόν η Γραμματεία θεωρεί πως καταπίπτει αυτή η τροπολογία αν εγκριθούν οι συμβιβαστικές 4 και 7. We will just, just give a second, colleague, to colleagues. Se posso, Presidente, l'emendamento... Anna Petrepete. Η τροπολογία 46 ζητά ψήφισμα, μάλλον μα θυμίζει ένα ψήφισμα που ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο το 2005 και εξάλλου αναφέρεται εδώ στα αρχικά εκτιμώντας ε, αποπειράται να επανυποβάλλει την υπόθεση της χρήσης ε, της διαφοροποιημένης ε, φορολογίας ε, για μεταβατικές περιόδους σε ορισμένες σε μειονεκτικές περιοχές. Αυτό δεν είναι αντίθετο με τα όσα αναφέρονται στην συμβιβαστική που ορίζει τις επενδύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη. Ας παραμείνει αυτός ο στόχος, αλλά στο στόχος θα μπορούσε να είναι και η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά και από τις φορολογικά έσοδα. Από πλευρά τη Γραμματεία δεν υπάρχει πρόβλημα να ψηφιστεί αυτή η τροπολογία. Αν από του πολιτικού ε, συντονιστέ δεν υπάρχει πρόβλημα για να ψηφίσουμε τη 46, μπορούμε να την ψηφίσουμε. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε για την τροπολογία 46. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Περνάμε στην συμβαστική 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. <coughs> Αποχέ, Εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 59 υπέρ. Α, συγγνώμη κύριος Λούχαν. Αναφέρομαι στην τροπολογία 59 που μιλά για την χορήγηση των κονδυλίων για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Κάνουμε μια συγκεκριμένη πρόταση, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τις τοπικές αρχές. Έτσι, οι περιφερειακές αρχές δεν θα χρειάζεται κάθε φορά να υποφέρουν από τις αλλαγές και κυβέρνησης που γίνονται τακτικά στις 27 χώρες μέλη. Η... Το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί και εγώ θα ήθελα να κάτω καταψηφιστεί η τροπολογία για να διατηρηθεί το άρθρο όσο είχε αρχικά. Και η πρόταση αυτή συμφωνία ανάμεσα στις περιφέρειες της κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Κομισιόν να παραμείνει ώστε οι επενδύσεις να είναι η προτεραιότητα. Ε, ζητώ από όλους τους συναδέλφους να καταψηφίσουν αυτή την τροπολογία. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ο κύριος Λούχαν έχει κάνει ένα σχόλιο σε σχέση με την τροπολογία 59 και από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν αίτημα της πολιτικής σας ομάδας, ήταν ένα γενικό σχόλιο για όλους τους συνάδελφους. Αφού ακούσαμε τον κύριο Λούχαν, πεσηφίζουμε για την τροπολογία 59. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε για την 59. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 ψήφοι υπέρ, 18 κατά. Πάμε στην τροπολογία 60. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 64 είχε αποσυρθεί. Πάμε στην 65 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω πρέπει να το ελέγξουμε. Ελέγχουμε για την 65 υπέρ, κατά και τα λοιπά, αλλά ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται 24 υπέρ 18 κατά. Πάμε στη συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Α, πάμε στην επόμενη σελίδα, συγγνώμη. 15. συμβεβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άμα κανείς δεν φωνάζει για έλεγχο, <laughs> εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 81. Ε, χωριστή ψηφοφορία. Έχουμε το πρώτο τμήμα της 81, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται κατά γνώμη μου. Τροπολογία 82, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 84. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86. Ε, Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 87. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 89. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ α συγγνώμη καταπίπτει καταπίπτει ναι 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99, 98 συγγνώμη, υπέρ, κατά, δεν ξέρω. Ελέγχουμε την 98. Κάποιες φορές σηκώνετε τα χέρια όταν έχω ήδη ρωτήσει πει κατά. 98, ελέγχουμε. Τέλος ψηφοφορίας, ναι. Υπέρ, 41 ε, υπέρ. 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ετολογία σκέψη 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στα εκτιμώντα. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7, τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, έλεγχος ηλεκτρονικός. Ελέγχουμε το εκτιμώντας ε, δέλτα τροπολογία 10. 24 κατά, καταπίπτει. Εκτιμώντας δέλτα τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω αλλά έχουμε για τη 12 Απορρίπτεται 26 προς 20. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 1 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στη ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης ηλεκτρονικά. Συνάδελφοι, άρχεται η ψηφοφορία υπέρ και κατά, αλλά ηλεκτρονικά. Ε, we can close the vote. It's 40 people are in favor, 5 against. 40 υπέρ, 5 κατά, μια αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν συγχαρητήρια στον εισηγητή. Now we move to point... Πάμε τώρα στο σημείο 9. Μάλλον θα πηγαίναμε στο 9, αλλά χθε συμφωνήσαμε με τους συντονιστές να α, αναβάλουμε τη ψηφορία. Πάμε στο 10 που είναι η έκθεση του Γιάννη Μπρεζίνα για τη διευκόλυνση του κλεισίματος διαφόρων ορυχείων. Η ε, κυρία Κρέλ, χθες που συντάξαμε την λίστα ψηφοφορίας, διαπιστώσαμε ότι ενδεχομένως η σειρά κατάθεσης ή μάλλον ψήφισης των ε, τροπολογιών 38, 39 και 40 ίσως πρέπει να αντιστραφεί. Διακόπτη η κυρία, διακόπτη η κυρία Χίπνερ. Για παρακαλώ ξαναπέστε γιατί δεν σας άκουσα. Νομίζω να αλλάξουμε, λέει η κυρία Κρέλ, την σειρά ψηφοφορία των τροπολογιών 38, 39 και 40. Να αρχίσουμε με την 40 και μετά να πάμε στην 38 και 39. Καλώς, καλώς φαίνεται ότι μόνο στη δική μου λίστα υπάρχει το σφάλμα αυτό. Δεν υπάρχει πρόβλημα λοιπόν. Η Πρόεδρος, ας αρχίσουμε και πρώτα η 21 έχει αποσυρθεί, 32 υπέρ. Έχω πολλές, πάρα πολλές. Μιλούμε. Διακόπτη Πρόεδρος. Έχει αποσυρθεί η 21, αυτό είπα στην αρχή. Αρχίζουμε λοιπόν με την 32. 32 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Αν θέλετε επαλήθευση μπορούμε να την κάνουμε. Όχι, καλώς. 33 υπέρ. Κατά. Ο ίδιος συσχετισμός δυνάμεων αποσύρεται. 18 ε, υπέρ. Κατά εγκρίνεται 35 υπέρ υπέρ λοιπόν κατά λυπούμε δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα η 35 παρακαλώ Α, θα την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την ψήφο αυτή. 35 λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Είναι σαφές ότι εγκρίνεται 34 προς 9. Συμβαστική τροπολογία 1 <clears throat> υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 38 εκπίπτει και 39 επίσης προχωρούμε 41 υπέρ κατά εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές Βλέπω του συντονιστέ και υποθέτω ότι του ακολουθείτε και ψηφίζετε υπέρ, αλλά δεν είναι σαφέ. Μην σηκώνουν μόνο τα χέρια τους οι, οι Λοιπόν, 43 υπέρ. Α, είναι ίδια. Είναι αυτό, αυτόσημη. Α, δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Καλά. 44 εκπίπτει, 20 εκπίπτει. Τι 20 λοιπόν. Την έχετε. Η συμβαστική 1 εγκρίθηκε. Άρα ψηφίζουμε την 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω λέει η πρόεδρος επαλήθευση αρχίζει πέρας 17 υπέρ 25 κατά απορρίπτεται 47 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 1. Μετιολογική σκέψη 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Ας κάνουμε επαλήθευση για την 2. Αρχίζει η ψηφοφορία. ...26 υπέρ, 17 κατά εγκρίνεται. 3. Ποιο είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία, τέλος ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία της. Who is against? Abstentions. This is against very... Αποχές. Ε, συγγνώμη, αλλά είναι οριακή ψηφορία. Θα πρέπει να γίνει λίγο λοιπόν επί του 4. Ψηφίζουμε. Πέρας. 24 υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο νούμερο 5, τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, σαφώς εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επίσης, 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 24 εδώ υπάρχει προφορική τροπολογία κόρτες, λάστρα όλοι Α, ε, υπάρχει κανείς που ενίσταται όχι, οκ, λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Αρχίζει η ψήφος. Πέρας. Απορρίπτεται. Με διαφορά δύο ψήφων. 20-22. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. 26 υπέρ 15 κατά. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. 16. Τροπογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται ας κάνουμε την επαλήθευση ωστόσο αρχίζει 19 υπέρ 25 κατά απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία τώρα, παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Αρχίζει. Πέρας. 39 ψηφί, υπέρ, 4 κατά και 2 αποχές. Εγκρίθηκε λοιπόν. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ και τη γραμματεία. Το σχέδιο γνωμόδοτησης Καμποβίνσκα για την αποδοτικότητα της ενέργειας στο σχετικό σχέδιο δράσης. Αρχίζουμε την ψηφοφορία με, τον, συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε την 10 λοιπόν. Αρχίζει η ψήφος. Πέρας. 25 κατά, άρα απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15, υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε την 15. Αρχίζει. Πέρας. 26 υπέρ, 15 κατά εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά αποχές σαφώς εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 16 υπέρ, κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται. Συμφωνείτε. Θέλει κανείς επαλήθευση. Καλώς. Επαληθεύουμε λοιπόν την 16. Πέρας. Σαφώς εγκρίνεται 27 υπέρ 16 κατά. Και η τελική ψηφοφορία ονομαστική με ηλεκτρονικό τρόπο. Πέρας. 42 υπέρ, καμία ψήφος κατά, δύο αποχές. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια. Τελειώσαμε τις ψηφοφορίες, αγαπητές και αγαπητοί. Όσοι εξημών επιθυμείτε να αποχωρήσετε, παρακαλώ, ησύχω. Προχωρούμε στο 12 της ημέρης της διαταξής. OG Βλάσακ European Urban Agenda και το μέλλον της στην περιφερειακή πολιτική. Το έχουμε μόνο στα αγγλικά το κείμενο όπως το γνωρίζετε. Θα δώσω το λόγο αμέσως ε, στον Όλτζι Βλάσακ για μια σύντομη ε, εισήγηση. Δεν πρόκειται να λάβουμε αποφάσεις σήμερα, ωστόσο το θέμα είναι σημαντικό. Ας αρχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση. Σας παρακαλώ λοιπόν, συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Όλτζι, έχετε το λόγο. Eh, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λέει ο κύριος Βλάσακ. Αν μου επιτρέπετε, θα κάνω μια εισήγηση σε σχέση με το έγγραφο το οποίο αφορά το μέλλον της πολιτικής ε, συνοχής καθώς και το ευρωπαϊκό αστικό περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε πάρα πολλά δεδομένα και από ό,τι φαίνεται οι πόλεις είναι πηγή ανάπτυξης. Μιλούμε για το 80% του ΑΕΠ στην Ευρώπη που εκπηγάζει από τις ε, αστικές περιοχές, το αστικό περιβάλλον. Έχουμε και για την αστική διάσταση μια προηγούμενη έκθεση. Η έκθεση αυτή πέρασε το 2009 και από τότε έχουν γίνει βέβαια διάφορες μεταβολές που έχουν επηρεάσει αυτή την πολιτική. Για να τα δούμε καλά τα πράγματα θα πρέπει πρώτα πρώτα να εξαρτάσουμε κάποιες έννοιες γιατί υπάρχουν ε, κάποιοι ειδικοί που παρόλα αυτά δεν χρησιμοποιούν τους σωστούς όρους και κυρίως η πολιτική. Άρα, πρώτα πρώτα θα πρέπει να έχουμε κάποιους ορισμούς. Τι θα πει πολιτική συνοχής, τι θα πει ευρωπαϊκό αστικό περιβάλλον. Τι εννοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά θα τα εντάξω στην ε, εισαγωγή το κείμενο μου. Επίσης, θα πρέπει να καλύψουμε εδώ κάποια νέα νομοθετήματα, κάποια νέα κείμενα, τα οποία τώρα τα επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Στατική Ενώση του 2020, την ε, πέμπτη έκθεση για την συνοχή, που είναι σημαντική και αυτή για το θέμα μας, οπότε και εγώ θα ήθελα να έχω τελειώσει τη δουλειά μου μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Και έτσι να μπορέσω να καλύψω όλα αυτά τα κείμενα στην εκθεσή μου και από της μεθοδολογίας θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να έχουμε συνεισφορά από διάφορους παράγοντες Θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε με μια μήνυα ακρόαση στην Επιτροπή μας. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για το έργο μου και συνεργαστήκαμε με διάφορους φορείς, ε, Eurocities, Telecities και άλλους. Γίναν κάποια εργαστήρια, κάποια σεμινάρια, οπότε είχα περισσότερη βοήθεια για να ξέρω ποιες είναι οι ανάγκες των πόλεων, τι περιμένουν από εμά. Ποια είναι τα προβλήματα, τι θέλουν επομένως και τελικά θα πρέπει όλα αυτά να συζητηθούν με όλους τους εμπλεκομένους. Θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή και με την Επιτροπή των Περιφερειών, που είναι η κυρίως αρμόδια. Επίσης θα πρέπει εδώ να εμπλακεί η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η Γενική Διεύθυνση για την Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής, αλλά βέβαια και η Επιτροπή, συγγνώμη και η ε, Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά με τους και οδησηγητές, αλλά και με άλλους συναδέλφους που τυχόν ενδιαφέρονται για το θέμα. Όπως προείπα, πέμπτη έκθεση για την συνοχή θα πρέπει να έχει αρχίσει να συζητείται μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Και θα αρχίσει επομένω μια ζήμωση, κάποιες επαφές όσον αφορά την πόλη του αύριο. Επίσης θα έχουμε και μια συνάντηση, ε, μάλλον συγγνώμη, η συνάντηση του Τολέδο θα φυγεί στα πλαίσια της έκθεσης αυτής και θα συζητηθεί. Άρα το πιο σωστό είναι να καλύψουμε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου των Υπουργών που έλαβε χώρα στην Λιέγη 23 και 24. Στην εισαγωγή επομένως θα περιλάβω κάποιους ορισμούς. Και Θέλω να καλύψω τα πιο σημαντικά ζητήματα, αυτά που ζητούν απαντήσεις. Αν έχετε κάποια συγκεκριμένη γνώμη, αν μπορείτε να με βοηθήσετε, αν έχετε κάποια ιδέα, ελάτε σε επαφή μαζί μου και πέστε μου. Επίσης, στην εισαγωγή, ίσως θα πρέπει να πούμε για το κατά πόσο χρειάζεται κάποιο είδου παρέμβαση από, από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώ μπορούμε να δαπάνε. άρα να δούμε σε ποιου τομεί μπορεί να παρέμβει η Ένωση. Και υπάρχει άλλο ένα τμήμα του κειμένου που ασχολείται με τις ε, ανάγκες σε τοπικό επίπεδο. Μιλούμε για έρευνα, για ερωτηματολόγια. Θα απευθυνθούμε στους εκπροσώπους των τοπικών φορέων. Ας πούμε, στον τσεχικό φορέα δήμων και κοινοτήτων. Γιατί υπάρχει κάποια σχετική έρευνα. Θεωρήθηκε ότι ωφέλησε πάρα πολύ. Είχαμε 650 ερωτήσεις που υπευλήθησαν και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Άρα θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι και οι ανάγκες των ευρωπαϊκών πόλεων. τι για την ευρωπαϊκή διάσταση και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους κοινοτικούς πόρους. Βεβαίως πάντοτε σεβόμενοι την επικουρικότητα. Τρίτο κείμενο, τρίτο τίτλο ή τρίτο τμήμα του κειμένου μάλλον θα είναι η εταιρική σχέση και η διακυβέρνηση. Εάν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα επίπεδα της πολυεπίπεδου διακυβέρνηση Όλα αυτά έχουν σημασία. Να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχουν περιθώρια για νέες πρωτοβουλίες. Εάν λαμβάνονται υπόψη σε κάθε επίπεδο ή κάθε ε, προτεραιότητα. Εάν μέχρι σήμερα έχει υπάρξει σωστή αντιμετώπιση. Επίσης, η αποκέντρωση των ε, διαρθρωτικών ταμείων που έχει επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα. Δούμε τι κινδυνοί υπάρχουν για να του αποφύγουμε. Σε αυτό το σημείο, αυτά τα θέματα θίγω, παρακάτω, ε, αν ασχολούμαι με την ανάθεση κάποιων αρμοδιοτήτων, κάτι το οποίο σήμερα γίνεται από πλευράς ε, δήμων στην ε, Ολλανδία. Και μάθαμε ότι αυτή η υπεργολαβία, αυτή η ανάθεση κάποιων θεμάτων λειτουργεί πάρα πολύ καλά στο Ρότερνταμ και αλλού. Τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά οι Ολλανδοί, οπότε θα πρέπει να δούμε αν αυτό το μοντέλο μας κάνει. Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι αρμοδιότητες θα υπάρχουν σε κάθε επίπεδο, περιφερειακό, τοπικό, ευρωπαϊκό, εθνικό. Και στο πρώτο τελευταίο τμήμα του κειμένου μου θα ασχολούμαι με τον συντονισμό των ενωσιακών πολιτικών. Υπάρχει ο πιο σωστός συντονισμός ή θα πρέπει να βελτιώσουμε και άλλα τα πράγματα. Θα βοηθηθούμε φυσικά από προηγούμενες εκθέσεις που έχουμε συνταχθεί. δούμε τώρα τι θα γίνει με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ή ολοκληρωμένο προγραμματισμό της στρατηγικής μας ή το στρατηγικό προγραμματισμό αν θέλετε γιατί θα πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τον προγραμματισμό το planning και αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί κατά τη γνώμη μου στο δε τελευταίο τμήμα του κειμένου θα ασχοληθώ με τον οικονομικό προγραμματισμό και την πρικοδότηση γιατί θα πρέπει να συζητηθούν τα γνωστά σχετικά προβλήματα. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν σημαντικά προβλήματα για την χρηματοδότηση των Δήμων. Οι Δήμοι θα πρέπει να συνάψουν δάνεια που σαν θέμα παρουσιάζει κάποια προβλήματα. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προσθέσουμε την όλη διαδικασία. Τους ελέγχους και την διαδίδαση κάποιων δεδομένων. Για να μην έχουμε επικαλύψεις ελέγχων. Γιατί επιβραδύνει τη διαδικασία των έχουμε επικαλύψει. Επίσης υπάρχουν και άλλα μέσα που διαθέσει μα, δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετά, κάποια χρηματοδοτικά μέσα τα οποία έχουμε διαθέσει μα και μπορούμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οπωσδήποτε και θέλω να ξέρω τη γνώμη σας για το πώς μπορούμε όλα αυτά να τα καλύψουμε. Αυτέ οι μερικέ ιδέε, συνάδελφοι. Ελπίζω να προκαλέσουν προβληματισμό, συζήτηση. Ε, όλα αυτά σας τα λέω σαν σύνοψη του τι θα έχω στον εγγραφό μου, οπότε και εγώ θα χαρώ να μάθω τις δικές σας ιδέες και προτάσεις. Έχουμε άλλωστε και μια συνάντηση εργασίας, όποιος την μπορεί να με βρει. Διότι θέλουμε πραγματικά με το κείμενο μας να βοηθήσουμε τους Δήμους. Χτες ο Γιώργος Γκούτμαν εξήγησε πώς έχουν τελευταίες εξελίξει όσον αφορά τους πόρους και την απορρόφηση αυτών. Πρέπει να κάνουμε ό,τι που περνάει από το χέρι μας για να τα πάμε καλά. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να προθυμοποιείται κανείς από τους ε, σκιώδεις ηγητές. Ρίκα Μάνερς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, τον εισηγητή για την θαυμασία έκθεση. Η προσέγγιση που επιλέγει είναι εξαιρετική. Ασφαλώς θα χρειαστούμε μια πολιτική για τα αστικά κέντρα. Σύμφωνο ότι η αφετηρία της εργασίας αυτής πρέπει να είναι οι ορισμοί. Ποια είναι τα αστικά κέντρα, ποιοι είναι οι χώροι των αστικών κέντρων, πώς ορίζονται. Ο αριθμός των πολιτών που κατοικούν εκεί είναι σημαντικός, κάποιο άλλο στοιχείο. Αυτά πρέπει να διευκρινιστούν. Από την άλλη μεριά πρέπει να λάβουμε υπόψη τα μητροπολιτικά κέντρα, όχι όμως μόνο τις μεγάλες πόλεις, αλλά και τις μικρές πόλεις και τις κόμες, γιατί και αυτές έχουν τα σχετικά προβλήματα. Πρέπει να προχωρήσει η εργασία αυτή σε στενή συνεργασία με άλλες πτυχές της πολιτικής συνοχής όπως της ανάπτυξης της υπαίθρου κλπ. Πρέπει λοιπόν να συναναπτυχθούν όλες αυτές οι πολιτικές μαζί με τις πολιτικές για τα αστικά κέντρα διότι βεβαίως υπάρχει διασύνδεση μεταξύ τους. Δεν θα πρέπει να αποφύγουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ των περιοχών αυτών. Γιατί αυτό δεν θα είναι προς το συμφέρον κανενός. Σε ό,τι αφορά την έκθεση, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τον τρόπο με τον οποίο ο συγητής αντιμετωπίζει τις διάφορες προκλήσεις. Από την άλλη μεριά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι μεταφορές παίζουν σημαντικό ρόλο. Και ιδίω οι οικολογικές ας πούμε μεταφορές, οι πράσινες μεταφορές πρέπει να ληφθούν πολύ περισσότερο υπόψη. Και η ευφύης ανάπτυξη αστικών κέντρων είναι επίσης πολύ σημαντική. Επίσης, πρέπει να μην λησμονούμε τους πολίτες που ζουν στα αστικά κέντρα. Πρέπει να συμμετάσχουν στην διαμόρφωση των πολιτικών. Ελπίζω αυτό να τονιστεί ιδιαίτερα στην τελική μορφή της εκθέσεως. Αυτή, αυτό το αίσθημα το συμμερίζεται η πολιτική μου ομάδα. Είναι σημαντική η πρόκληση λοιπόν της ανάπτυξης των αστικών κέντρων και υποστηρίζουμε την προσέγγιση του εισηγητού. Κύριε Καρυμαντελή. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Ε, επιμένω τώρα πρώτα στον κρίσιμο ρόλο των πόλεων, των αστικών κέντρων και για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Ε, τα έχω ξαναπεί αυτά την προηγούμενη φορά. Αλλά τρία τέταρτα των καυσαερίων προέρχονται από τα αστικά κέντρα. 80% της ενέργειας καταναλώνεται στις πόλεις. Πρέπει λοιπόν αυτά τα πράγματα να πούμε ξεκάθαρα, διότι ο αγώνας για την διατήρηση του κλίματος θα παιχτεί στις πόλεις. Έτσι λοιπόν βιώσιμες πόλεις θα πρέπει να είναι η πρόκληση του αιώνα για να διατηρηθεί η πόλη και να ωφελήσει και η φύση βέβαια και να ωφελήσει τις μελλοντικές γενιές. Δεύτερο, οι μεγάλες αποκλίσεις μέσα στις ίδιες τις πόλεις. Οι μεγάλες ανισότητες. Σήμερα οι ευρωπαϊκές πόλεις διαθέτουν βεβαίως πλεονεκτήματα, συγκεντρώνουν τον πλούτο, τον πολιτιστικό πλούτο, τον οικονομικό πλούτο και ούτω καθεξής, αλλά ο μεγαλύτερος αριθμός των ευρωπαϊκών πόλεων αντιμετωπίζουν και σημαντικότατες κοινωνικές ε, ανισορροπίες. Φτώχεια, έλλειψη παιδείας, ε, κακή ποιότητα στέγη, κακή ποιότητα περιβάλλοντος. Αυτά είναι πραγματικότητε, είναι συγκεκριμένε πραγματικότητες για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. Εδώ λοιπόν εντοπίζεται μια άλλη πρόκληση που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων αφενός θα έχουμε πόλεις ανταγωνιστικές, αφετέρου θα έχουμε πόλεις οι οποίες θα εγκαταληφθούν στην παρακμή. Δεν επιτρέπεται όμως να έχουμε ευρωπαϊκές πόλεις δύο ταχυτήτων. Γι' αυτό και πρέπει να εγκρίνουμε, την, να στερεώσουμε καλά την ε, ημερήσια διάταξη αυτή, την ατζέντα mm. για τις πόλεις και οι πόλεις να ενταχθούν μέσα στην περιφερειακή ανάπτυξη. Να εμπνευστούμε δε από τα επιτυχημένα πειράματα για παράδειγμα, την κοινοτική πρωτοβουλία Urban. Η επιτυχία των πολιτικών για τις ε, πόλεις με συμμετοχή όλων των φορέων, τοπικών, περιφερειακών και άλλων, να φτιάξει μια πολιτική συνοχής με συμμετοχή των πόλεων. Όπως για παράδειγμα έγινε με την συνθήκη των ε, δημάρχων που συνυπέραψαν 1.700 δήμαρχοι το πρόγραμμα Urban λειτουργήσε. Γιατί δεν ξεκινούμε ένα παρόμοιο πρόγραμμα Urban για την ενέργεια. Θυμίζω εξάλλου τον συμβιβασμό που προέκυψε από τον τριμερή διάλογο του κ. Έτιγκερ κυρίως 146 εκατομμύρια ευρώ που θα βοηθήσουν στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στις πόλεις. Το πρόγραμμα, το, συγγνώμη, το Ταμείο ΦΕΝΤΕΡ μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια των ευρωπαϊκών πόλεων ώστε να υιοθετήσουν προγράμματα υπέρ του κλίματος, να ε, αφιερωθεί δηλαδή και στην διαχείριση των προγραμμάτων με μια ενεργό εταιρική σχέση των τοπικών φορέων για να προχωρήσουν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις για την ενέργεια και για την στέγη. Εν τέλει, θα υπενθυμίσω ότι είπε ο κύριος Ντελμπάρ, πρόεδρος του ΚΟΤΕΡ των ε, περιφερειών. η πόλη δεν θέλουν να ζητείτε απλώς η γνώμη τους. Αυτό είπε. Θέλουν να μπουν στην συμπαραγωγή της πολιτικής συνοχής. Αυτό το στοιχείο πρέπει να περιληφθεί στην έκθεση. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και βεβαίως θα συμμετάσχω στην εκπόνηση της εκθεσής σας. Κύριε Βλασάκ, ευχαριστώ. Φραντσέσκο Ντε Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο συνάδελφο Κοτσολίνο δεν μπορεί να συμμετέχει στη συζήτηση λόγω ανελημμένων θεσμικών υποχρεώσεων στην Ιταλία. Ε, είναι σκιώδη συζητητή για αυτό το έγγραφο εργασία. Γι' αυτό Θα ήθελα να σας μεταφέρω την ε, συμβολή του και την εκτίμησή του για αυτό το έγγραφο και για τον ε, ρόλο της πολιτικής συνοχής. Επί της ουσίας. Σημεριζόμαστε τις αρχές που εκφράζονται στο έγγραφο, κυρίως όσον αφορά την αναγνώριση του ρόλου κλειδιού που παίζουν οι πόλεις για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Όσον αφορά το περιεχόμενο του εγγράφου, Είμαστε υπέρ των μηχανισμών ε, εξουσιοδότησης ε, που βασίζεται σε μια διακυβέρνηση πολυεπίπεδη και ωστόσο αυτές οι έννοιες δεν είναι τελείως νέες. Στον προγραμματισμό 2007-2013 ήταν ήδη δυνατόν να αναθέσουμε ορισμένες αρμοδιότητες στις τοπικές αρχές ε, ως ενδιάμεσους οργανισμούς ο τοπικός λοιπόν προγραμματισμός θα έπρεπε να ενταχθεί μέσα στα περιφερειακά προγράμματα και να αποτελέσει μάλιστα ένα απόσπαστο τμήμα τους. Μια ρυθμίση, ρύθμιση η οποία ωστόσο εκτός από σποραδικές περιπτώσεις έχει μείνει μόνο στα χαρτιά. Πριν να προτείνουμε λοιπόν ένα ανάλογο μοντέλο διακυβέρνησης, θα ήταν καλό να καταλάβουμε ποιε είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν στην ανάθεση του προγραμματισμού και στην εφαρμογή προγραμμάτων που έχουν ενταχθεί στο ευρύτερο περιφερειακό πρόγραμμα αλλά με βάση τις τοπικές αρχές. Αυτό θα πρέπει να γίνει ε, και κυρίως να εμπλακούν οι πόλεις από την αρχή του προγραμματισμού στο πρόγραμμα. Δύο παρατηρήσεις επιπλέον. Ε, καταρχήν ε, μια εισαγωγική παρατήρηση για το ρόλο που μπορεί να έχει η αστική ανάπτυξη για την ανά, υπέρβαση των δυσκολιών, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τώρα οι μετροπολιτικές περιοχές, να δούμε πώς μπορούν να αποτελέσουν ένα πραγματικό κίνητρο, κινητήρα μάλλον για την ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα ακριβώς στις μεγάλες αστικές ε, περιφέρειες έχουν γίνει πιστητότερα ε, ο αντίκτυπος της κρίσης, αλλά και έχει επιδεινωθεί η περιβαλλοντική κατάσταση. Γι' αυτό και θα πρέπει να δώσουμε σε αυτούς τους στόχους ε, στην στρατηγική 2020. Θα πρέπει δηλαδή οι πόλεις να αποτελέσουν το επίκεντρο των ε, τομεακών περιφερειακών που εσωματώνουν την πολιτική, την κοινωνική, την πολιτική, την οικονομική και ε, την περιβαλλοντική. Μια πραγματική δηλαδή και βιώσιμη ανάπτυξη ώστε να δοθεί και πάλι στις αστικές περιοχές ε, ο κεντρικός χαρακτήρας που τους αξίζει. Άρα λοιπόν η συνεργασία μας με τον εισηγητή, τον κύριο Βλάσλακ, τον οποίο ευχαριστώ για την δουλειά που έχει κάνει και κυρίως για τη δέσμευσή του να δώσει μια αναπαντελεσματική απάντηση σε ένα πρόβλημα και σε ένα ζήτημα εξαιρετικά ε, ευαίσθητο λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα η κυρία Ερμήνια Ματσόνη, ναι, σκιώδης για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου για τη δουλειά του και συναδέλφου Βλάζακα και κυρίως να τον ευχαριστήσω για την ανοιχτή πρόσκληση σε εμπλοκή πραγματική και σοβαρή των σκιωδών εισηγητών. Εκτιμώ ιδιαίτερα τον, την μέθοδο συμμετοχής και την οποία ακολούθησε ο κύριος Βλάζακ και την ε, ε, χρησιμοποίησε και σήμερα το πρωί. Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία μας στη φάση επεξεργασίας του κειμένου, έτσι ώστε να μην υπάρχουν στη συνέχεια διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς που ε, να παρεμβαίνουν ε, σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Οι αστικές περιοχές έχουν μεγάλη σημασία και είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνουμε. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει πως θα πρέπει να ξεχνάμε κάποιες ε, ασφαλιστικέ δικλείδε και την γνώση επί τη οποία έχουμε παγιώσει την ε, Ευρώπη. Ο εισηγητή ξεκινά από μια σωστή παραπομπή στην έκθεση για την αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής στη νέα προγραμματική περίοδο. Σε αυτήν αναφέρομαι και εγώ. Γιατί είναι σωστό να σκεφτούμε το βάρος που έχουν οι αστικές περιοχές, οι πόλεις στην Ευρώπη. 80% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει στις πόλεις και στις περιφέρειές τους και παράγουν το 70 με το 80% του εγχώριου ακαθάριστου προϊόντος. Οι αστικές περιοχές είναι ο μεγαλύτερος κινητήρας ανάπτυξης της οικονομίας μας ξεκινώντας από το βασικό κύτταρο που είναι οι μικρές ε, και μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συζητήσαμε χθε και που αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό. Σχεδόν ε, είναι η απόλυτη πλειοψηφία των, ε, του επιχειρηματικού μας ιστού. Πρέπει ωστόσο να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει μια αστικοποίηση, μια αστιφιλία, ε, νέα, ένα νέο κύμα αστιφιλίας ε, που οδηγεί σε διάφορα περιβαλλοντικά προϊόντα, ε, περιβαλλοντικά συγγνώμη, προβλήματα, αλλά οδηγεί και σε μια επιδίνωση της ποιότητας ζωής στα κέντρα τα αστικά. Πολλές φορές γίνεται αναφορά στην ανάγκη διατήρησης της ευκαιρίας μιας ανά, της δυνατότητας μιας συνεργασίας ανάμεσα στις ε, αστικές περιοχές και στις περιοχές της υπαίθρου, ώστε να υπάρξει ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη. Μέσα σε αυτή τη λογική καθίστανται στόχοι προτεραιότητας, η αύξηση της αντιπροσώπευσης των πληθυσμών που ζουν στις πόλεις ε, σήμερα, που δεν αντιπροσωπεύονται αρκετά στα διάφορα προγράμματα. Θα πρέπει δηλαδή να αναλάβουμε και να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα, ενώ ταυτόχρονα να διατηρήσουμε και την θετική εμπειρία του mainstreaming που έχει χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα Urban μέσω της ενίσχυσης των ολοκληρωμένων διαδικασιών και της ε, προσέγγισης της ανωδικής, από κάτω προς τα πάνω και κατά την άποψή μου θα πρέπει να αφήσουμε μέσα στο πλαίσιο αυτής της εργασίας ολοκλήρωσης αυτών των προσπαθειών μας της ανάπτυξης των αστικών περιοχών να μην μπερδευτούμε με μια δύσκολη, έναν δύσκολο ορισμό των αστικών περιοχών που νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το αναλάβουν τα κράτη. Με τη βάση λοιπόν αυτών των σκέψεων, εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις για το κείμενο του συναδέλφου, για τον ορισμό του πλαισίου, δηλαδή την περίμετρο μέσα στην οποία θα πρέπει να λειτουργήσει αυτή η αστική ατζέντα. Εγώ δεν νομίζω πως είναι περιοριστικό στις εισαγωγές της αστικής ε, ατζέντα στην πολιτική την περιφερειακή, αλλά είναι κάτι φυσιολογικό όσον αφορά το μέσο urban είναι μια στιγμή αξιοποίησης ε, του εργαλείου αυτού. Πιστεύω πως ε, η αναμπλοκ οργάνωση του κειμένου θεωρούμε πως είναι αρμονική και πλήρης Ίσως ε, εγώ θα ήθελα να περικόψω λίγο τα σημεία 3 και 4 και τα 6 και 7. Όπως ήδη είπα, για τις αστικές περιοχές ίσως θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε την αναφορά στην ε, ταξινόμηση όξ που ισχύει τώρα και που έχει δώσει θετικά αποτελέσματα. Πιστεύω ότι για την αναγνώριση των προτεραιοτήτων θα ήταν σωστό και υπό το φως των παρεμβάσεων που άκουσα από τον συνάδελφο Ντεάντζελης θα ήταν ίσως σκόπιμο να κάνουμε έναν απαρίθμηση των κατευθύνσεων της στρατηγικής 2020 που μας δείχνουν το δρόμο για μια ευφύ Ευρώπη αλλά και βιώσιμη και αντί να μιλάμε για smart growth, να μιλάμε και για ανάπτυξη και ε, βιώσιμη και για όλους. Τώρα, η ανάθεση διαφόρων αρμοδιοτήτων είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι και αυτό ένα μέσο το οποίο ήδη έχουμε πειραματιστεί, έχουμε ήδη δοκιμάσει και προβλέπεται. Απλώς πρέπει να προσέξουμε ώστε να τοποθετηθεί σε ένα, ένα αρμονικό πλαίσιο που θα σέβεται την αρχή της διακυβέρνησης της πολυεπίπεδης. Τώρα όσον αφορά την πρόταση ενός διατομιακού συντονισμού, είμαι πεπισμένη πως αυτός είναι ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, διότι σε σχέση με την λογική της ολοκληρωμένης προσέγγισης που πρέπει να στηρίξουμε και που θα πρέπει να μας δώσει και θετικά αποτελέσματα. Τέλος, ε, είναι αυτονόητο ότι συμμερίζομαι όλες τις προσπάθειες που θα γίνουν για να απλοποιηθούν οι διαδικασίες η ε, κυρίως όσον αφορά τις δραστηριότητε των τοπικών αρχών που πολλές φορές ε, οδηγεί σε πολύ μεγάλο φόρτο και που παρεμποδίζει την παραγωγικότητα των μέσων που εμείς θέτουμε στη διάθεση των περιφερειών. Αυτή είναι μια καλή βάση λοιπόν, επί της οποίας μπορούμε να δουλέψουμε. Επανεπιβεβαιώνω την εκτίμησή μου για την πρόσκληση που μας έκανε ο εισηγητής για μια συμμετοχή από πλευρά των σκιωδών εισηγητών και σίγουρα εγώ θα συμμετέχω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Λάμπερτ Φανίστελ Ρόι. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος γιατί είναι καλό το έγγραφο. Επίσης συμμετείχα στην ακρόαση που διοργανώθηκε Πράγμα το οποίο με οδηγεί στο να θέσω ορισμένα ερωτήματα. Καταρχήν τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, ε, ε όπως το κάναμε από το Urban, ε, μη πρέπει να αρκούν τα εργαλεία που έχουμε. Πρέπει να συμπληρώσουμε όπως κάναμε το Airban. πρέπει να δούμε με βάση την, την στατηγική του 2020, πρέπει να προβλέψουμε νέα μέσα. Δεν θέλουμε μόνο να δίνουμε επιδοτήσεις και ε, βοήθεια. Θα πρέπει οι επενδύσεις νέου τύπου να είναι δυνατές και μάλιστα να βρεθεί ένας κοινός παρανομαστής ανάμεσα στις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Θα πρέπει να συμβάλλουμε δηλαδή στις επενδύσεις και να βασιστούμε στην βιωσιμότητα των ε, διαφόρων περιοχών και των πόλεων το Ταμείο Συνοχής θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε εν μέρη, αλλά θα πρέπει αυτό να το ενισχύσουμε στην έκθεση, να είμαστε υπέρ του κοινοτικού προγράμματος, όπως έγινε με το ε, Όρμπαν, είτε υπέρ μιας άλλης προσέγγισης. Θα πρέπει κάπου να γίνει μια επιλογή και πιστεύω ότι ο κύριος Βλάζακ μετά από τα αποτελέσματα της ακρόασης ε, ε, ε, ασχολήθηκε πολύ με το θέμα και γι' αυτό και τον καλό να προβεί σε επιλογές. Και η Ένωση της Καινοτομίας είναι ένα, μία από αυτές τις πρωτοβουλίες ε, τις ε, εμβληματικές. Μας είπαν ότι ένα από τα βασικά θέματα είναι οι έξυπνες πόλεις, όχι μόνο πιο πράσινες πόλεις, αλλά οι βιώσιμες μια ματιά ή να τονίσει αυτές τις πρωτοβουλιες τις εμβληματικες μας ειπαν οτι ενα απο τα βασικα θεματα ειναι οι εξυπνες πολεις οχι μονο πιο πρασινες πολεις αλλα οι βιωσιμες και εξυπνες πολεις οι πολεις ισως λοιπον αυτη η εκθεση θα πρεπει να ριξει μια ματια η να τονισει αυτες τις δράσεις που θέλουμε να κάνουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. και τα λοιπά συμφωνώ με τα όσα είπε η κυρία Μαντζόνη. Köszönöm a szót, tisztelt eh, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Megpróbálok nagyon röviden fogalmazni. Először is. Τελευταίο από τον κύριο Σεγγέντη. Σα ευχαριστώ. Θα, είμαι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον κύριο Φλάσσα για το εξαιρετικό του έγγραφο. Υπάρχουν δύο πράγματα ωστόσο που πιστεύω πω λείπουν από αυτό το έγγραφο, αλλά φυσικά αυτό είναι δική μου άποψη. Νομίζω πως πρέπει να διαφοροποιήσουμε ανάμεσα στις πόλεις στην Δυτική Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη. Από το πρώην Συμβούλιο Αμοιβέ Οικονομικής Συνδρομής. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα της οικογένειάς μου. Η οικογένειά μου δουλεύει στους αγρούς και εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Και το 1950 οι κομμουνιστές πήραν τα χωράφια, τα ζώα, τα μηχανήματα και τα πάντα και χρειάστηκε να πάνε στην πόλη. Εγώ μεγάλωσα στην πόλη λοιπόν. Στην Ανατολική Ευρώπη λοιπόν υπάρχει αυτή η, στη, Δυτική συγγνώμη, Ευρώπη η δημιουργία των μεγάλων αστικών κέντρων ήταν μια φυσική πορεία ενώ στην Ανατολική Ευρώπη ήταν καταναγκαστική και πρέπει να γίνει αυτή η διαφοροποίηση. Κάτι ακόμα το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην έκθεση αυτή είναι η εναρμόνιση του ρόλου των ε, αστικών και των ε, γεωργικών περιοχών. Ακούσαμε ότι το 80% του ΑΕΠ ε, παραγωγείται στις πόλεις. Ξεχνάμε όμως την, την ανθρώπινη πλευρά. Οι πόλεις είναι αβίωτες. Πρέπει να σεβαστούμε την άποψη των ανθρώπων των πόλεων. Πρέπει να ενδιαφερθούμε για αυτούς. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε το περιβάλλον, την ρήπανση, ο κύριος ε, Φανίστερ το ανέφερε αυτό, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται μόνο να έχουμε πράσινες πόλεις, αλλά ευφυείς πόλεις, ούτως ώστε να μπορούν να είναι βιώσιμες και ανεκτές και στο μέλλον. Θα πρέπει να μιλήσουμε για την έλλειψη υγιεινής διατροφής έχουμε τεράστιες, ε, τεράστιους πόρους διατροφικούς αλλά όχι υγιεινούς πόρους. Αυτό ισχύει για τη Δυτική Ευρώπη. Και έπειτα οι εθνοτικές συγκρούσεις είναι παρούσες στις πόλεις. Στην Δυτική Ευρώπη οι μετανάστες προκαλούν το πρόβλημα. Στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ουγγαρία είναι οι Ρώμα που δημιουργούν το πρόβλημα. Θα πρέπει αυτά τα προβλήματα να τα, να τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε κάνει λόγο για την ανάπτυξη των πόλεων και την ανάπτυξη από οικονομική άποψη, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και τους ανθρώπους που θέλουν να απομακρυνθούν από τις πόλεις αλλά δεν μπορούν να το πράξουν γιατί είναι αδύνατον να ζήσει κανείς ζώντα σε μια ε, αγροτική περιοχή. Γι' αυτό και η ανάπτυξη υπαίθρου είναι πολύ σημαντική. Όταν σκεφτόμαστε την περαιτέρω ανάπτυξη των πόλεων θα πρέπει να έχουμε και να στηρίξουμε και τα μικρά ε, χωριά και κομοπόλεις και να αναπτύξουμε την Ήπεθρο. Δεν θα πρέπει μόνο να μιλάμε για συμβολικές χειρονομίες προς τις ε, περιοχές της Ήπεθρου, θα πρέπει να προβούμε σε πραγματική δράση, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης στα μικρά χωριά και στις ε, περιοχές της Ήπεθρου, να υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης. Σε ένα μικρό χωριό θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή απαραίτητη υποδομή. Ο κόσμος που ζει στις πόλεις αλλά στα προάστια θα πρέπει επίσης να μπορεί να έχει πρόσβαση στην πόλη. Για να συνοψίσω για να βοηθήσω τους δυτικούς συναδέλφους να καταλάβουν, θα πρέπει να ε, μιλήσουμε για τις διαφορές, να δούμε τις διαφορές, όχι να χωρίσουμε τις πόλεις από την Ήπεθρο, α, το αντίθετο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για την έκθεση του κυρίου Βλάσε και ελπίζω Όζη να μην χρειάζεται να πάρει το λόγο. Να επαναλάβω ότι καλή όλους... Άντε, ένα λεπτό, ένα λεπτό γιατί έχουμε αργήσει. Ένα λεπτό. Μισό λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το μόνο πράγμα που θέλω να πω ότι πολλά από αυτά που αναφέρθηκαν εδώ Είναι πράγματα που δεν τα ανέφερα επίτηδες. Είχαμε μιλήσει για τις δημόσιες μεταφορές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε προηγούμενες ε, ευκαιρίες και θα σας δώσω τα έγγραφα που έχουμε από την ακρόαση για τις ευφύς πόλεις. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν ήδη καλυφθεί. Θα σας τα ξαναστείλω και θα το συμπεριλάβω και στην έκθεσή μου. Τώρα όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές και το περιβάλλον στις πόλεις, συμφωνώ πως είναι τεράστιο το ζήτημα και ότι είναι κάτι που, θα, που έχουμε λάβει υπόψη, διότι ενδιαφερόμαστε για περισσότερη δουλειά στον τομέα και για περισσότερη στήριξη. Λάβαμε λοιπόν την ε, τεκμηρίωση και θα το συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Τώρα για την Ήπεθρο. Φυσικά και δεν πρέπει να στήσουμε σύνορα ανάμεσα στις πόλεις και την Ήπεθρο. Όχι, αυτοί που ζουν στην Ήπεθρο κοντά στις πόλεις ε, πρέπει να είναι περήφανοι για τις πόλεις τους και αντιστρόφως ανάλογα. Αλλά η συνεργασία θα πρέπει να είναι πιο ουσιαστική. Θα πρέπει λοιπόν όλες αυτές οι στρατηγικές καθώς και οι περιφερειακοί, να συνδυαστούν. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και προσβλέπω στη μελλοντική μας συνεργασία. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να σας πω ένα σοβαρό αίτημα. Εχθέ αποφασίσαμε να αλλάξουμε την ατζέντα, ώστε να καταστεί δυνατό ο κύριος Ντεάντζελης να παρουσιάσει την έκθεσή του. Γιατί έχει τρένο να πάρει σύντομα. Ε, την εξετάσουμε δηλαδή πριν από το διάλειμμα. Δηλαδή τώρα έχουμε τρεις εκθέσεις για μια ώρα σημαίνει 20 λεπτά την έκθεση. Αν δεν τα κάνουμε αυτά, τότε δεν μπορώ να δεχτώ το αίτημα του κ. Ντεάντζελης και θα πρέπει να πανέλθουμε στην προηγούμενη ημερήσια διάταξη. Σας παρακαλώ λοιπόν, πολύ σύντομε παρουσιάσεις επί της ουσίας για να διατηρήσουμε την ατζέντα ως έχει. Χισμένοβα, έκθεση Χισμένοβα. Τώρα να σας θυμίσω τελευταία φορά κάναμε έκθεση για το θέμα και η κυρία Χισμένοβα δεν θεώρησε να, απαραίτητο να κάνει περαιτέρω σχόλια. Γι' αυτό θα προβούμε κατευθείαν στη συζήτηση. Αν χρειάζεται λοιπόν να συνεχίσουμε τη συζήτηση, είστε πρόσδεκτοι, αλλά παρακαλώ λάβετε υπόψη το γεγονός ότι δεν έχουμε χρόνο. χρόνο. Δεν έχουμε... Από ό,τι κατάλαβα η κυρία Ισμένοβα δεν θέλει να κάνει μια ακόμα εισήγηση μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην συζήτηση αν, στο, με τους κοιόδης εισηγητές, αν κάποιοι από εσάς θέλετε να πάρετε το λόγο. Μετά από τη συζήτηση του περασμένου μήνα. Η Σαμπίν Θα είμαι σύντομη. Ευχαριστώ και πάλι για την συνεργασία με την κυρία Χισμένοβα. Οι συζητήσεις ήταν πολύ χρήσιμες υπενθυμίζω τα δύο θέματα που είχα θίξει και την προηγούμενη φορά. Δεν υπάρχει λόγος ούτε χώρος να επιβαρύνουμε με πολυγλωσία όλες τις τοπικές ή περιφερειακές αρχές. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα σημείο, μία αρχή, η οποία να μπορεί να τους προσφέρει τις ε, πληροφορίες που χρειάζονται στη γλώσσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Τα αγγλικά ούτως ή άλλως θα είναι ε, διαθέσιμα και ίσως και η γλώσσα μιας ακόμη χώρας. Όχι όμως πολλές γλώσσες εργασίας. Ευχαριστώ που τηρήσατε τον ε, χρόνο. Γκάιερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Συνήθως οι συνεδριάσεις των Επιτροπών όπου είμαι τακτικό μέλος συμπίπτουν με τις δική σας. Πάντως χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Είμαι σκιώδης για την ανταλλαγή αυτή απόψεων, για την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών, για την πολυγλωσία δεν είμαι βέβαιος εάν με την προσέγγιση που έχουμε επιλέξει μπορώ να είμαι σύμφωνος. Μήπως δηλαδή τελικά με την γνωμοδότηση αυτή κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά παρά καλό. Διότι θα αρχίσουν ατελείωτες συζητήσεις για τα αγγλικά, για την ανάγκη να προσθεθούν και άλλες γλώσσες, γλώσσες συγγνώμη, θα πρέπει πολύ απλά η ίδια η τοπική ή η περιφερειακή αρχή να αποφασίσει που θα ρίξει το βάρος εάν δηλαδή είναι χρήσιμο η αυτή να προσελκύσει κάποιους προσφέροντας και άλλη μια γλώσσα. Η πολυγλωσία άλλωστε υπερβαίνει και τα όρια της αρμοδιότητας της Επιτροπής. Έχω ορισμένες τροπολογίες υπόψη, τις οποίες θα υποβάλω για την έκθεση της κυρίας Ισμένοβα σχετικά με το ποιες εγγυήσεις πρέπει να εξασφαλίσουμε μέσα στην οδηγία παροχής υπηρεσιών, ώστε τελικά να ωφελεί περισσότερο η οδηγία αυτή παρά να προκαλεί ζημία. Διότι έχουμε δει στην Γερμανία περιπτώσεις όπου το πλεονέκτημα, δηλαδή η ανάπτυξη της ελευθερίας στην ενιαία αγορά, στην ουσία μειώθηκε από τον φόβο του κοινού αν θα διατηρηθεί η δυνατότητα επιλογής υπηρεσιών, ποιος θα είναι ο ρόλος των αστικών κέντρων, τα συζητήσαμε και πριν αυτά, εάν θα προκύψει ανταγωνισμός, τι γίνεται με την ασφάλεια των κεκτημένων των εργαζομένων, και από πλευράς παρόχων υπηρεσιών, για παράδειγμα για ε, τοπικές κοινότητες αυτή η αρχή που λέει ίση αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο τόπο πρέπει να ισχύσει σε όλη την Ευρώπη. Οι δεμοί άνθρωποι τρομάζουν από αυτή την απελευθέρωση που βλέπουν και την μείωση των κοινωνικών προδιαγραφών. Ας μην μας εκπλήσει τότε όταν μειώνεται το ενδιαφέρον και ο του κοινού υπέρ της Ευρώπης. Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι να υπάρχει ένα συνομιλητής στην ε, τοπική αρχή για τους εργαζόμενους. Και νομίζω επίσης ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε περισσότερο τις τοπικές κοινότητες και δήμους. Αλλά να περιορίζονται στην παροχή των υπηρεσιών εκείνων που ωφελούν πραγματικά τους πολίτες. Σας ευχαριστώ. Κύριε Χισπένοβα, θέλετε να λάβετε πάλι τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το γεγονός ότι οι σκιώδεις συζητητές συνεισφέρουν με πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Η κυρία Βερχάιν έκανε την πρόταση που περιλαμβάνεται στην παραγραφό 4 για την αρχή της πολυγλωσίας... στις ε, διάφορες, στα διάφορα contact points και η ενθάρρυνση προς τις χώρες μέλη να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία από τις κοινοτικές γλώσσες ώστε να διασφαλίζεται μια ταχύτητα ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερομένων και της αρχής. Στην αρχική μου πρόταση Είχα υποβάλει το στοιχείο αυτό. Η κυρία Βερχάιν συμμετέσχε στις αρχικές μας συζητήσεις και την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Επίσης, ευχαριστώ τον κύριο Γκάιερ, σκιολυσιγητή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θα περιλάβω τις προτάσεις που έγιναν στο κείμενό μου και ελπίζω όταν θα ανοίξει η διαδικασία για την υποβολή νέων προτάσεων να μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα ολοκληρωμένο κείμενο που εν τέλει νομίζω θα είναι πραγματικά χρήσιμο για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Αναμένω λοιπόν τις προτάσεις των συναδέλφων μου και είμαι βεβαία ότι το κείμενο που θα προκύψει εν τέλει θα είναι πολύ χρήσιμο. Η πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 9η Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Αυτό θα μας επιτρέψει να ψηφίσουμε στην τελευταία μας συνεδρίαση 30 Νοεμβρίου, δηλαδή 1η Δεκεμβρίου. Έτσι λοιπόν 9 Νοεμβρίου 6 το απόγευμα. Τώρα, το υπαριθμό 17 της σημερινής διάταξης, σχέδιο γνωμοδότησης De Angelis, η βιομηχανική ανάπτυξη στην παγκοσμιοποιημένη εποχή. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων, δεν καλούμαστε να λάβουμε αποφάσεις. Κύριε <coughs> De Angelis, λαμβάνετε το λόγο και μην λησμονείτε ότι έχουμε ακόμα την κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ναι, και ζητώ συγγνώμη που ζήτησα πιο νωρί να συζητηθεί το θέμα. Θα είμαι πολύ σύντομο. Έκανε καλά η Ευρώπη που τόνισε το θέμα του βιομηχανικού μέλλοντος και το κάνουμε αυτό σε μια στιγμή ιδιαίτερη δυσκολίας και κρίσης που πλήττει πάρα πολλές επιχειρήσεις, ένα σωρό εργαζόμενους και πάρα πολλές οικογένειες. Και αυτό το κάνουμε με στόχο να βγούμε από την κρίση και να αναζωογονήσουμε την ανάπτυξη, την ανάκαμψη και κυρίως την ανταγωνιστικότητα του ε, βιομηχανικού μας συστήματος. Όσον αφορά λοιπόν τις εργασίες αυτής της Επιτροπής ε, και ε, μετά από μια επαφή που είχα σήμερα αυτή την εβδομάδα με τους υπόλοιπους ηγητές, ε, τους κοιόδους ηγητές και τους ευχαριστώ μάλιστα για την συνεργασία τους, θα ήθελα Ε, να σας παρουσιάσω πολύ πολύ σύντομα τις απόψεις. Είναι προφανώς ότι κάθε βιομηχανική πολιτική θα πρέπει καταρχήν να είναι συνεπής με τους γενικούς στόχους που ορίζει η Ευρώπη σε ε, αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών, δηλαδή με σεβασμό των ε, ε, ανταγωνιστικών στάνταρ ε, και προδιαγραφών με τις υπόλοιπες παγκόσμιες αγορές και κυρίως όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες ε, συζητήσαμε χθε και για το ρόλο τους στην πολιτική συνοχή αντιπροσωπεύουν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Θεωρώ λοιπόν πως μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανάκαμψη των ευρωπαϊκών βιομηχανιών δεν μπορεί να ξεχνά την τις μικροεπιχειρήσεις τις, και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρξει ένας επικοδομητικός διάλογος με τους φορείς της αγοράς και απέναντι και στους ε, εργαζόμενους να είμαστε πιο ε, δυναμικά, να μιλήσουμε για το Small Business Act και για μια ευρωπαϊκή στρατηγική πρόσβαση στην πίστοση. Άλλο σημαντικό θέμα είναι ε, το θέμα των κέντρων αριστείας ως ε, μοχλών ανάπτυξης ε, μέσα στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς ε, κύκλους και τα κέντρα κατάρτισης. Σε σχέση τέλος ανάμεσα στον παραγωγικό κόσμο και τα επανεπιστήμια, κυρίως για την ανάπτυξη ζωγόνηση ενός ε, ε, ανθρώπινου δυναμικού που λείπει σήμερα και που είναι απαραίτητο για τη συγκεκριμένη στήριξη της ζωής των επιχειρήσεών μας. Να επενδύσουμε λοιπόν στην καινοτομία, στην έρευνα, στην αριστεία για να ευνοήσουμε την ανάκαμψη και την ανάπτυξη. Τέλος, να επιβεβαιώσουμε και πάλι το θέμα της ε, κεντρικού ρόλου των τοπικών αρχών, των περιφερειών και των, της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα μέσω των, του Ευρωπαϊκού του Κοινωνικού Ταμείου, του Πλαισίου για την Ανάπτυξη και την Ανταγωνιστικότητα, καθώ και για τη νέα συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτά θα πρέπει να είναι οι διάβλη μέσω των οποίων οι τοπικές αρχές και οι περιφερειακές αρχές θα μπορέσουν να επιβεβαιώσουν και πάλι τον κεντρικό τους ρόλο. Εύχομαι αυτά τα μέσα όχι μόνο να επιβεβαιωθούν και να συνεχιστούν μετά το 2013, αλλά και ότι θα υπάρχει μεταξύ τους μεγαλύτερη εναρμόνιση και περισσότερα κονδύλια που είναι απαραίτητα για τις ε, κατευθύνσεις αυτές που είπαμε για να εγγυηθούμε την ανάπτυξη και την απασχόληση. So... Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές η ε, κυρία Μάντερ. Ε, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εισήγηση αυτή ήταν εξαιρετική. Και βεβαίως και οι σκιώδεις εισηγητές ε, κλήθησαν να συμμετέχουν εξ αρχής. Έχω εγώ τέσσερις παρατηρήσεις να αναφέρω. Καταρχήν, στο σύνολο του είναι σημαντικό το μέτρο αυτό γιατί οι παραδοσιακές βιομηχανικές ζώνες περνούν μια μεταβατική περίοδο με μεγάλες δεκιμάσεις όσον αφορά την απασχόληση γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στη, στα νέα κοιτάσματα, κοιτάσματα απασχόλησης. Να τονίσω λοιπόν την λειτουργία των ε, ε, κλάστερ των κέντρων δηλαδή των βιομηχανικών ε, έτσι ώστε η παραγωγή να είναι συγκεντρωμένη, να υπάρχει μια υποδομή που θα διευκολύνει πολλές επιχειρήσεις μαζί. Ε, είναι πολύ σημαντικό η εκμετάλλευση των, φυσικών πόρων να γίνεται με βιώσιμο τρόπο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη σημασία τους για το σύνολο της κάθε περιφέρειας και έπειτα για τις κλιματικές αλλαγές. Ε, είναι σημαντικό οι κλιματικές αλλαγές να μην θεωρηθούν μόνο απειλή για κάθε ζώνη, αλλά και ως μια ευκαιρία ιδιαίτερα για τις ε, ειδικές, ε, την, την ειδική ανάπτυξη και τέλος για τις περιφερειακές ε, ε, τις πιο απομακρυσμένες δηλαδή περιοχές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε των ανταγωνιστικότητας και υποδομών. Αυτά ήθελα να σας πω εν συντομία. Σας ευχαριστώ. Η συνεργασία ήταν πολύ καλή μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, δεν βλέπω άλλο να θέλει να πάρει το λόγο. Η κυρία μαντάλης δεν είστε σκιώδης. Εσείς αντικαθιστάτε κάποιον. Μάλιστα. Merci, euh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντεάντζελη, καταρχήν να σας ζητήσω συγγνώμη εξ του συναδέλφου κυρίας ε, Κατρίν Γκρές που δεν μπορούσε να είναι παρούσα αλλά που ήθελα να σας μεταφέρει τις απόψεις της για το γνωμοδότησή σας. Το κείμενό σας ε, παίρνει προσανατολισμούς για τους οποίους σας είχε μιλήσει και η κυρία Γκρέσ και άρα είναι ευτυχής γι' αυτό. Μιλάμε για ε, για την στήριξη των πιο αδύναμων περιφερειών, να αντιμετωπίσουν τις ε, οι πιο ευαίσθητες περιοχές την παγκοσμιοποίηση χρειάζονται βοήθεια και αναφέρονται και οι, οι περιφερειακές ε, περιοχές, ε, δηλαδή οι πιο απομακρυσμένες που συχνά τις ξεχνάμε. Ε, σας ευχαριστούμε λοιπόν για την δουλειά που κάνατε μέχρι τώρα. Δυστυχώς όμως δεν αναφέρατε την ε, μετακίνηση της οικονομίας και των παραγωγικών κύκλων γιατί από το πλαίσιο της κρίσης μία από τις λύσεις είναι η ανάπτυξη τοπική. Αν θέλουμε βιώσιμες θέσεις που να μην μπορούν να μετακινηθούν, αυτές, ε, αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Επίσης λυπούμεθα που δεν αναφέρατε, δεν υπογραμμίζεται ο ρόλος των περιφερειών στην οικολογική μετατροπή των, των ε, βιομηχανιών. Θα πρέπει λοιπόν να τονιστεί αυτό και να το χρηματοδοτηθούν μη ε, λέμαριες σε ενέργεια βιομηχανίες που δεν ρηπαίνουν. Θα πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε για τα των κλιματικών αλλαγών και να αντικαταστήσουμε τις ε, την ενέργεια από τα αστερά καύσιμα. Υπάρχουν ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, μεταφορέ πολύ πιο καθαρέ και ούτω καθεξή. Τέλο, η περιφέρεια θα πρέπει να παίξει ρόλο στην συνοδεία των τομέων που βρίσκονται σε ύφεση. Η αυτοκινητοβιομηχανία ή η αεροναυπηγική. Θα πρέπει να στηρίξουμε την αναμετατροπή της τεχνογνωσίας των εργαζομένων χρηματοδοτώντας ε, σχέδια κατάρτιση γιατί έτσι θα μπορέσουν να ε, καταρτιστούν εκ νέου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ρόζα Ισταράς Φεραγκούτ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βασικά θέλω να πω ότι η γνωμοδότηση του εισηγητή είναι πολύ ισορροπημένη και είναι προφανές γιατί υπάρχει μεγαλύτερη συνένεση από ότι αντιφάσεις. Το ίδιο δίνει σημασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο εισηγητής αλλά και στη συνογή 99% των επιχειρήσεων ε, είναι μικρομεσαίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν το μεγαλύτερο δημιουργό θέσεων απασχόλησης σύμφωνα με τα στοιχεία του 2009. Είμαστε σε κρίσιμη συγκυρία και αυτό λέει και ο συγητή και επομένω θα πρέπει αυτή η κρίση να μα κάνει να ενεργήσουμε με ρυθμού ε, κατεπήγοντο και επομένω γι' αυτό θα πρέπει να κατεβάσουμε ένα κατεπήγοντο όσον αφορά τη μαύρη οικονομία, όσον αφορά όσα δεν δηλώνονται, ούτω ώστε να προσέχουμε μια που βρισκόμαστε σε κρίση για αυτέ όλε τι δραστηριότητε. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο αφορά ε, τι περιφερειακέ, ε, τι περιφέρειε, συγγνώμη, τι νησιωτικέ και ένα άλλο κομμάτι το οποίο αφορά την πολιτική του τουρισμού, την βιομηχανία του τουρισμού και έτσι θα τονίσουμε το πόσο σημαντικός είναι και αυτός ο κλάδος ε, μια που πρόκειται για τον πρώτο τουριστικό προορισμό και πρόκειται για τις Βαλιαρίδες όπου η ατιμομηχανή της οικονομίας είναι ακριβώς ο τουρισμός. Και να δούμε πώς ε, θα, θα μπορέσει να, να ανατονώσει τον τουρισμό η, η Κομισιόν με τα μέτρα της και οπότε ελπίζουμε ότι με τη συμβολή μας αυτή θα βελτιώσουμε το κείμενο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε εμείς, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελε κάποιος άλλος να μιλήσει. Ιδάλλως, τότε θα ξαναγυρίσουμε στον εισηγητή, κύριε Ντιάντζελες. Μήπως θέλετε να συνοψίζετε. Και ευχαριστώ πολύ σύντομα. Με λαβή της παρατηρήσεις και τις ενδείξεις των συναδέλφων για βελτίωση του κειμένου, κυρίως ορισμένα σημεία όπως το θέμα του κεντρικού χαρακτήρα των περιφερειών, την χρήση των πόρων, το θέμα της γνώσης, της καινοτομίας της έρευνας, των κέντρων, των κλάστερ. Νομίζω πως θα κάνουμε μια πολύ σημαντική δουλειά σε μια πολύ ε, ευαίσθητη περίοδο για την οικονομία της Ευρώπης. Εμείς ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος, και έτσι ε, ολοκληρώνουμε τα του σημείου αυτού. Η δε κατελτική προθεσμία θα είναι στις 9 Δεκάτου, στις 6 το απόγευμα, ούτως ώστε να μπορέσουμε γέρος να εγκρίνουμε την έκθεση πριν ε, αρχίσει να ασχολείται η Ήτρε με αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Επομένως, 9 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα κλείνει η προθεσμία για τις τροπολογίες. Τώρα θα ήθελα να πάμε στο σημείο υπαριθμών 14. Κρέλ. Θα πρέπει να ε, έρθει. Έρχεται, να την τώρα μόλις. Έρχεται η κυρία Κωνσταντς Κρέλ. Θα πρέπει να σας πω, αν δεν συμμετέχετε στην Επιτροπή ΣΟΥΡ, ε, εντάξει όλοι συμμετέχουν σε αυτή την ειδική επιτροπή, ούτως ώστε να αποκρισταλωθεί η θέση του Κοινοβουλίου για τις δημοσιονομικές προοπτικές και ξέρετε ότι αυτή η επιτροπή έχει εντολή μέχρι τον Ιούνιο του 2011. Όμως θα είμαστε μέχρι τότε έτοιμοι, θα έχουμε τελική θέση του Κοινοβουλίου και πρόκειται να γίνει τον Ιούνιο ακριβώς η ψήφιση του σχετικού κειμένου. Και η Επιτροπή ΣΟΥΡ ασχολείται και τώρα συζητεί και επεξεργάζεται θέματα οριζόντιας φύσης για τις δημοσιομικές προοπτικές αλλά περ' τον Ιανουάριο θα αρχίσει να ασχολείται με τα πιο κλαδικά ζητήματα της επιμέρους πολιτικές και για αυτό η, η γνωμοδότηση της δικής μας Επιτροπής θα έχει ιδιαίτερη σημασία και τώρα θα δώσουμε τη σκητάλη στην Κωνσταντς Κρέλ η οποία επεξεργάζεται το έγγραφο που αφορά την συμβολή της δικής μας Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Μόλις έρχομαι τώρα από την Επιτροπή ΣΟΥΡ, διαπιστώνω κατ' επανάληψη ότι εκεί τουλάχιστον κάθε δεύτερος ομιλητής μιλεί περί πολιτικής συνοχής. Και αυτά τα πρόσωπα δεν ήταν ούτε είναι μέλη της ε, Περιφερειακής Επιτροπής. Άρα το θέμα του απασχολεί πολύ. Ε, πρόκειται και για πολλά χρήματα. Βέβαια, νομίζω πρέπει να συντάξουμε μια στεναρή, ας πω έτσι, γνωμοδότηση, ξεκάθαρη, για να μπορέσει να αντέξει και στις διάφορες αμφισβητήσεις που θα έλθουν και από την Επιτροπή αυτή αλλά και στην Ολομέλεια. Όπως είχαμε πει, είχα ελπίσει μάλιστα ότι θα είχαμε περισσότερο χρόνο για την γνωμοδότηση, έχοντας ωστόσο μιλήσει με την πρόεδρο της Επιτροπής ΣΟΥΡ, κυρία Χάουκ, μου δημιουργείται η εντύπωση ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το αργότερο μέχρι τέλη Ιανουαρίου να έχουμε ψηφίσει και εγκρίνει την γνωμοδότηση, Ώστε ο εισηγητή του τη ΣΟΥΡ, κ. Γκαρίγα, να μπορέσει να την εντάξει, τη γνωμοδότησή μα δηλαδή, στην έκθεσή του. Να μην έρθουμε δηλαδή εκ των υστέρων και ίσια ίσια να την ξεφυλίσουν για να δουν αν κάτι τους ενδιαφέρει να περιλάβουν. Έτσι, για τους επόμενους δυόμιση μήνες το χρονοδιάγραμμά μας θα πρέπει να είναι πολύ σφιχτό και για το λόγο αυτό στην συνεδρίασή μας του Δεκεμβρίου θα υποβάλω το σχέδιο της γνωμοδότησης. Ελπίζω πριν από αυτό το χρονικό σημείο να έχω λάβει από τις πολιτικές ομάδες σχόλια και προτάσεις. Εισαγωγικά θα πω τώρα το εξής. Νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε πολλά θέματα στην γνωμοδότηση. Τεχνικά όμως, δυστυχώς, έχουμε τους γνωστούς περιορισμούς στα, στην έκταση των κειμένων των γνωμοδοτήσεων. Θα μπορέσω λοιπόν να περιλάβω διάφορα πράγματα, αλλά με πολύ σύντομο τρόπο. Εγώ ίδια θα υποβάλω τροπολογίες, ώστε να καταστήσω μέσω των τροπολογιών αυτών πιο σαφή τα όσα θα θέλω να πω. Παράδειγμα, θεωρώ σωστό να συζητήσουμε μέσα στη γνωμοδότηση για τις προτεραιότητες που θέλουμε. Στο σχέδιο της γνωμοδότησης, για παράδειγμα, μπορεί να θέλω να πω ότι πρέπει να ενισχύσουμε την έρευνα αυτό ωστόσο χρειάζεται μια αιτιολόγηση, μια θεμελίωση. Αυτό θα το κάνω ασφαλώς μέσω μιας τροπολογίας. Για το θέμα τώρα, για το κυρίως θέμα, ελπίζω να με βοηθήσουν οι συνάδελφοι, γνωρίζοντάς μου τις θέσεις τους σχετικά με το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί. Γνωρίζετε ότι η πολιτική συνοχής στην παρούσα δημοσιονομική πρόπτικη έχει 384 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό. Η πολιτική συνοχής θεμελιώνεται ρητά μέσα στην συνθήκη της Λισαβόνας, πολύ πιο ξεκάθαρα. Συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν και η περιφερειακή συνοχή. Θα έχουμε σε μεγάλα μέρη αυτής δικαίωμα συναπόφασης, και για τη στρατηγική 2020 η πολιτική συνοχής παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Σήμερα στην Επιτροπή ΣΟΥΡ μας επιβλήθη έγγραφο. Θα είναι σημαντικό δε αυτό για τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό μετά από το 2013. Για την ώρα έχουμε 123 εκατομμύρια δηλαδή 1% του ΑΕΠ θα πρέπει να είναι δισεκατομμύρια αυτό το ποσό ε, ε, για τα 500 εκατομμύρια των 500 ε, εκατομμύρια των πολιτών δαπανάτε επομένως ανά και κατά κεφαλή 246 ευρώ για να εξασφαλιστούν όλα ειρήνη, ευημερία, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικό μοντέλο, που το κοινωνικό μας μοντέλο είναι βέβαια ασύγκριτο με οποιαδήποτε άλλο στον κόσμο, για να μπορούν να σπουδάσουν, για να μπορούν να μετακινηθούν, για να μπορούν να διακινηθούν, να μπορούν να εγκατασταθούν όπου θέλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αναπτυχθεί μια ενιαία αγορά και για να γίνουν προσπάθειες υπέρ των εργαζόμενων και των καταναλωτών ξαναλέω το ποσόν 246 ευρώ κατά κεφαλήν τον χρόνο. Δηλαδή στην ουσία τίποτα. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί στην αρχή του κειμένου μας. Όταν λέμε ότι θέλουμε πολιτική συνοχή μετά το 2013, η οποία να διαθέτει και προϋπολογισμό που να είναι επαρκής. Αν θέλουμε να μπούμε στη στρατηγική 2020 Ωραία είναι όλα αυτά. Αλλά στις τρεις κατηγορίες Smart, Sustainable, Εφής, Αϊφόρος και ποιο είναι το άλλο δεν θυμάμαι τώρα. Μπαίνουμε στην τρίτη κατηγορία. Αλλά η πολιτική συνοχής δεν είναι ταυτόχρονα και μέρος μιας πολιτικής smart, μιας ευφυούς, ευφυούς πολιτικής, καθώς επίσης μιας βιώσιμης πολιτικής. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε, διότι εκεί αρχίζει, από εκεί, αρχίζει από είναι η αφετηρία γιατί εκεί διαγράφεται ο κίνδυνος να πούν κάποιοι προτιμούμε μια ευφυή πολιτική ή προτιμούμε μια βιώσιμη πολιτική και άρα μπορούμε να μειώσουμε τα ποσά που δίνονται στην πολιτική συνοχή και τονίζουμε περισσότερο κάποια άλλα. Αυτό πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα ποσοστά δηλαδή που χρειαζόμαστε στην πολιτική συνοχή για την ανάπτυξη και έρευνα, για την προστασία του κλίματο, για την αποδοτικότητα τη ενέργεια είναι σαφώ μεγαλύτερα από τα επιμέρου προγράμματα που έχουμε στη διάθεσή μα μέσα στον κοινωτικό προπολογισμό και που εγώ δεν θέλω να αλλάξω διότι η πολιτική συνοχή στην περίπτωση αυτή είναι πολιτική υπέρ των περιφερειών. Από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να προχωρούμε σε τομεοποίηση μένουν οι περιφέρειες απ' έξω. Και νομίζω ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στις περιφέρειες, ώστε αυτές οι περιφέρειες να μπορούν να αποφασίζουν πώς θα διαχειριστούν τα χρήματα που του διατίθενται και πρέπει να λεχθεί καθαρά στις χώρε μέλη, καθώς επίσης βέβαια και στις περιφέρειες, ότι δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί και μάλιστα μέσα σε περίοδο κρίσης να αποφασίσουν να κάνουν εξοικονομήσεις και να θεωρούν τότε ότι οι περιφέρειες μπορούν ίσως από άλλες πηγές, από εθνικές πηγές να ε, αντλήσουν χρήματα για να κάνουν περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτά Πρέπει να τα καταστήσουμε σαφή στη γνωμοδότησή μας. Εξετάζοντας τώρα πώς διαμορφώνεται η πολιτική συνοχής στις 273 περιφέρειες που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε στόχους 1, ε, περιφέρειες δηλαδή του στόχου 1, του στόχου 2, αλλά με τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωστάτου του 2007 ο χάρτης έχει αλλάξει. Θα κοιτάξω να βρω και τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία. Αλλά έχουμε τον χάρτη του 2007 όπως είπα που καθιστά σαφές ότι ο αριθμός των περιφερειών στόχου 1 θα μειωθεί σημαντικά από το 2013 και μετά και θα μετακινηθεί σαφώς προς τις νέες χώρες μέλη. Κάτι το οποίο θα έχει ως συνέπεια, εάν υποχωρήσουμε στις πιέσεις ορισμένων χωρών μελών και συγκεντρώσουμε τα κονδύλια κυρίως σε περιοχές στόχου 1, αυτό λοιπόν θα σημαίνει τότε ότι μεγάλα τμήματα τη παλαιά Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα λαμβάνουν πλέον ουδέμια χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχή. Αλλά αυτό θίγει όχι μόνο παλαιέ χώρε μέλη, αλλά και νέε χώρε μέλη. Χώρε όπω η Μάλτα, η Σλοβενία. Και με τα στοιχεία του 2007 θα μείνουν απ' έξω. Στην γνωμοδότησή μα λοιπόν πρέπει να καταστεί σαφέ ότι όταν μιλούμε για τις υφιστάμενες κατηγορίες, περιοχές στόχου 1 και στόχου 2. Χρειαζόμαστε να έχουμε στόχου, περιοχές στόχου 1, στόχου 1 και στόχου 2 που να μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική συνοχή. Γιατί η πολιτική συνοχή δεν σημαίνει μοναχά ενίσχυση των μειονεκτικών περιοχών, σημαίνει επίσης καταπολέμηση των προβλημάτων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαίνει προσπάθεια μείωσης των μεγάλων ανισοτήτων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μονάχα πρέπει να αυξηθεί η ενίσχυση που δίνεται σε ένα τμήμα. Πρέπει να υπάρξει μια συνολική ανάπτυξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μου φαίνεται αναγκαίο και από οικονομική άποψη αλλά και από κοινωνική. Και όσοι λένε ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί παρά να κινείται προς μία μόνο κατεύθυνση, αυτό είναι λάθος. Η αλληλεγγύη πρέπει να κινείται προς διάφορες κατευθύνσεις και αμοιβαία. Εάν εξετάσουμε ποιες προτεραιότητες επιθυμούμε να υποστηρίξουμε, στο ψήφισμά μας που εγκρίναμε πρόσφατα είπαμε ορισμένα πράγματα και νομίζω ότι αυτό είναι και το ελάχιστο που θα πρέπει να περιλάβουμε στη γνωμοδότησή μας. Πρώτιστα λοιπόν αηφόρο οικονομική ανάπτυξη με ευεργετικές επιδράσεις στην αγορά εργασίας, καλύτερη και περισσότερη απασχόληση. Αυτό πρέπει να είναι βέβαια η πρώτη στη προτεραιότητα, σύγχρονη υποδομή, υποδομή και στον τομέα των μεταφορών, αλλά και στην υδροδότηση, στην αποχέτευση, στις επικοινωνίες μέχρι και στην ενέργεια. Αυτά όλα μπορούν να ενταχθούν υπό τον τίτλο «Υποδομές». Να μπουν όλα αυτά εκεί. Ασφαλώς οι ανάγκες εν προκειμένου των νέων χωρών μελών είναι μεγαλύτερες. Για τις παλές χώρες μέλη θα δούμε αν μπορούμε να σκεφτούμε και εδώ στην Επιτροπή μας, εάν δηλαδή πούμε περισσότερο Ταμείο Συνοχής για την υποστήριξη των υποδομών ή να πούμε όχι ας γίνουν οι ενισχύσεις υποδομών από το Περιφερειακό Ταμείο. Αυτό πρέπει να το δούμε και στην πρόταση που θα κάνουμε στην Επιτροπή ΣΟΥΡ. Άλλη προτεραιότητα που νομίζω κανείς δεν αμφισβητεί είναι ο τομέας έρευνα, καινοτομία, ανάπτυξη τεχνολογίας που να είναι κοντά στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Η μεταφορά δηλαδή των πορισμάτων της έρευνας Άρα υποστήριξη κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες από μόνες τους δεν είναι σε θέση να κάνουν έρευνα. Και αυτό νομίζω πρέπει να είναι από τα κύρια θέματα. Και ε, βλέποντας τα υπό το πρίσμα της περιφερειακής πολιτικής τα πράγματα αυτά, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι σημαντικό να κρίνεται στις ίδιες τις περιφέρειες ποιες κατευθύνσεις θα λαμβάνονται προς τα που θα δίνονται οι διάφορες ενισχύσεις. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από το πρόγραμμα στήριξης για την έρευνα, όπου είναι διαφορετική και πρέπει να είναι διαφορετική η νοοτροπία, διότι εκεί πρέπει να γίνονται πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν μόνες τους οι χώρες μέλη. Είναι λοιπόν διαφορετική αφιτερία από αυτό που λέμε προκειμένου, ότι θέλουμε δηλαδή μέσα στις ίδιες τις περιφέρειες να στηρίξουμε την έρευνα και την καινοτομία. Σε σχέση τώρα λοιπόν με αυτό το θέμα, για μας θα είναι σημαντικό να θέσουμε θέματα παιδείας, ξεκινώντας από την σχολική εκπαίδευση. Χωρίς να μπούμε στις αρμοδιότητες των χωρών μελών, σύμφωνοι, αλλά να δώσουμε υποστήριξη σε μια προσπάθεια βελτίωσης της σχολικής εκπαίδευσης. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις τάσεις που ήδη διαγράφονται στην παρούσα περίοδο. Σχολική εκπαίδευση, παραπέρα εκπαίδευση. Μη λησμονούμε βεβαίως και την δημογραφική εξέλιξη, κατάρτιση διαβίου που πρέπει να τεθεί πολύ εντονότερα μέσα στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής, διότι νομίζω ότι είναι και σημαντικός παράγοντας που θα εξασφαλίσει την παραμονή των βιομηχανιών στους τόπους όπου βρίσκονται. Και αυτό έχει και σχέση με, το, με την κοινωνική διάσταση της πολιτικής συνοχής. Γιατί έτσι θα μας επιτρέψει να καταπολεμήσουμε την φτώχεια, δημιουργώντας προγράμματα που θα επιτρέψουν την ένταξη στην αγορά εργασίας. Αυτά για μένα είναι και η πραγματική θεμελίωση του κοινωνικού ταμείου μέσα στην πολιτική συνοχής ή τέλος πάντων υπό την αιγίδα της. πρέπει να επιμείνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελεί και πρέπει να παραμείνει μέρος της πολιτικής συνοχής. Δεν πρέπει να φύγει από εκεί. Να του δοθεί μεγαλύτερη ορατότητα, να συμμετάσχουν περισσότερο όλες οι περιφέρειες, να παραμείνει όμως μέσα στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Το ίδιο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε και για την Ήπεθρο. το Ταμείο δηλαδή για την Ανάπτυξη της Υπέθρου να παραμείνει ή να ενταχθεί κάτω από την αιγίδα της πολιτικής συνοχής. Αυτό θα έχει πράγματι και δημοσιονομικές επιπτώσεις, διότι αν κάνουμε σωστό συνδυασμό μπορούμε μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου να διαμορφώσουμε πιο αποτελεσματικά κάποια πράγματα, να κάνουμε και κάποιες εξοικονομήσεις για παράδειγμα αναθέτοντα ορισμένα πράγματα, ορισμένα προγράμματα στο Ταμείο Ανάπτυξη τη Υπέθρου. Εκεί χρειάζεται λοιπόν κάποια ευκαμψία την οποία πρέπει να δείξουμε και στις διαπραγματεύσει για τον προϋπολογισμό μετά το 2013. Εν προκειμένου, αν ε, γίνουμε πιο αποδοτικοί και στην ανάπτυξη της Υπέθρου, πιο αποτελεσματικοί, θα δούμε αν μπορούμε να πούμε ότι ρίχνουμε το βάρος του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου στην ανάπτυξη του αστικού κέντρου και της περιφερειάς του, γιατί μας ενδιαφέρει να προωθήσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη στην πόλη και στο περιβάλλον της, που να έχει και οικονομική και κοινωνική διάσταση. Και εδώ υπάρχει δυνατότητα λοιπόν να δαπανηθούν χρήματα με τρόπο πολύ αποτελεσματικότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Ένα, μια άλλη, όχι ακόμα τελευταία, αλλά πραγματικά πάρα πολύ σημαντική προτεραιότητα είναι η εξή. Ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ταχθούμε υπέρ της διαμεθοριακή συνεργασίας υπό τις διάφορες μορφές που έχει, όχι μονάχα τη διαμεθοριακή συνεργασία, έχουμε την συνεργασία περιφερειών, έχουμε την συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών, έχουμε τις μακροπεριφέρειες. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα εντάξουμε και μέσα στον προπολογισμό. Να δώσουμε δηλαδή μεγαλύτερη βαρύτητα, αφού στην πραγματικότητα έχει αποδειχτεί ότι η περιφερειακή πολιτική και από μόνη της προσφέρει ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία. Η περιφερειακή πολιτική που θα ενισχύσει αυτήν την διαμεθοριακή συνεργασία καθίσταται ορατή, ακόμα πιο ορατή ως προστιθέμενη αξία. Και το μόλις 2,5% που δίνεται στην διαμεθοριακή συνεργασία, πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε αν μπορούμε να αυξήσουμε το ποσοστό αυτό. Και θα πρέπει να σκεφτούμε βέβαια ταυτόχρονα πόσο θα προχωρήσουμε. Αν δηλαδή στην γνωμοδότηση θέλουμε πράγματι να ταχθούμε ή μάλλον να εκφράσουμε καθαρά πώς θέλουμε εμείς να δούμε τον προϋπολογισμό. Ασφαλώς με κανένα τρόπο δεν πρέπει να δεχθούμε να είναι μικρότερος από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Ξεκινώντας από τα 350 δις εκατομμύρια ευρώ, να δούμε τι γίνεται με την προσαρμογή στις τρέχουσες τιμές κτλ. Με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει ο υπολογισμός, ώστε εγώ δεν ξέρω ποια μορφή θα λάβει τελικά ο προπολογισμό, αλλά αναλογικά δεν πρέπει να γίνει μικρότερος. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε να παραμείνει στα επίπεδα που έχουμε μέχρι τώρα. Χρειαζόμαστε λοιπόν για να επιτευχθεί αυτό ευφυεί προτάσεις. Θα προτείνω στην παρούσα επιτροπή να κάνουμε προτάσεις σχετικά και με το τι θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται πλέον να χρηματοδοτηθεί. Είμαι, αναμένω με ανυπομονησία να δω εάν υπάρχουν κάποιες ιδέες που θα λέγουν ότι κάποια πράγματα που χρηματοδοτούνται τώρα από την πολιτική συνοχή μπορούν ίσως στο μέλλον να οργανωθούν καλύτερα στο εθνικό επίπεδο. Πρέπει να δούμε λοιπόν εάν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Σας ομολογώ ότι μέχρι τώρα δεν μου έρθε καμία ιδέα σχετικά. Ίσως όμως οι συνάδελφοί μου να έχουν κάτι να πούν σχετικά. Κάτι που πρέπει να καταστήσουμε σαφές και το είπα ήδη στην αρχή της ομιλίας μου είναι ότι δεν θέλουμε το ομοιοποίηση του προϋπολογισμού. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό. Αν και βέβαια στην πολιτική συνοχής και για λόγους δημοσιονομικούς πρέπει να το πούμε και στην γνωμοδότηση Ασφαλώς και πρέπει να λάβουμε υπόψη τις προκλήσεις της αλλαγής του κλίματος, της δημογραφικής αλλαγής, πρέπει να ληφθούν υπόψη και να τεθούν ως προτάσεις. Ιδέες κυκλοφορούν πολλές για διάφορα πράγματα. Γνωρίζετε ότι πολλοί ενδιαφέρονται να δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο μεταφορών εγώ το βλέπω αυτό με ιδιαίτερη επιφύλαξη γιατί πιστεύω ότι μπορεί να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτά σχετικά με τις προτεραιότητες. Στη γνωμοδότηση θα πρέπει να πούμε κάτι και για την διάρκεια της επόμενης δημοσιονομικής πρόπτικης. Κατά τη γνώμη μου και υπάρχουν διάφοροι λόγοι που συνηγορούν υπέρ της ιδέας μιας επταετίας και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια σχεδιασμού για τις χώρες μέλη και τις περιφέρειες και σε ό,τι αφορά για την αντιμετώπιση των διαφόρων αντιδράσεων, διότι κάποιες μακροοικονομικές διαδικασίες χρειάζονται κάποια χρόνια για να εκδηλωθούν. Επίσης, ορισμένα προγράμματα για να προχωρήσουν. Τα 7 χρόνια μου φαίνεται ότι είναι λοιπόν μια καλή πρόταση. Υπάρχει και μια πρόταση που λέει 2 φορές 5, δηλαδή συνολικά μια δεκαετία έχω ορισμένες αμφιβολίες εάν αυτή η σκέψη ότι θα πρέπει δηλαδή μετά την πρώτη πενταετία να γίνει μια ενδιάμεση ε, επανεξέταση μήπως οδηγήσει αυτό πολλούς να πιστέψουν ότι δεν είναι ε, ο, καθορισμένος ο προϋπολογισμός για όλο το διάστημα αλλά μετά την πάροδο της πρώτης πενταετίας θα πρέπει να γίνει αναθεώρησή του. Οπότε, εάν εξ αντιθέτου δεν γίνει τέτοια αναθεώρηση μετά την πρώτη πενταετία, τότε βέβαια αυτομάτω τα 2 επί 5 σημαίνει 10 και 10 χρόνια είναι υπερβολικά μακρύ χρόνο και δεν επιτρέπει κάποια ευκαμψία. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, νομίζω ότι 7 χρόνια είναι μια χρυσή μεσιόδο. Θα πρέπει να περιλάβουμε κάτι και για τους κανόνες και τη διαχείριση του Ταμείου Συνοχής, απλοί ξεκάθαροι κανόνες που να εναρμονίζονται όσο είναι δυνατόν και με τα άλλα μεγάλα προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω άκουσα άλλιστα πριν από λίγο, γιατί στην Επιτροπή ΣΟΥΡ επανέρχονται στην ιδέα ότι θα μπορούσε να γίνει και 100% χρηματοδότηση ορισμένων έργων. Εγώ νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι δεν είναι σωστή αυτή η ιδέα και ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η συγχρηματοδότηση. Θυμάμαι παλαιότερα την διαρθρωτική πολιτική με εκείνο το 100% που ήταν στην ουσία δωρεάν χρήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προέκυψαν έργα τα οποία είχαν, δεν είχαν καθόλου ε, βιώσιμο χαρακτήρα, ήταν στην ουσία περιτά με λίγα λόγια, φτιάξανε γέφυρες πάνω από ποτάμια που δεν υπήρχαν. Να σα το πω έτσι. Η συγχρηματοδότηση είναι σημαντική διότι εξασφαλίζει και το ότι υπάρχει πράγματι κάποιο συμφέρον της περιφέρειας να προωθήσει ένα έργο. Και όταν βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς όπως την παρούσα οικονομική κρίση και η συγχρηματοδότηση είναι δύσκολο να γίνει από ορισμένους τοπικούς φορείς να εξετάσουμε εάν ίσως μπορεί να υπάρχει κάποια ευκαμψία από μέρος μας υπό ορισμένε συνθήκες και όρους. Επίσης, να τοποθετηθούμε σχετικά με το ποια ποιοι δημοσιονομικοί μηχανισμοί θα πρέπει να εντάσσονται στην ε, πολιτική συνοχή στο μέλλον. Για την ώρα γίνονται μόνο επιχορηγήσεις, να δούμε εάν ίσως μπορούν να δοθούν δάνεια ε, με εκείνα τα ανακυκλούμενα ταμεία για να επιτυγχάνεται περισσότερη αποτελεσματικότητα. Ρίχνω μια στιγμή μια ματιά και στο ρολόι, θα σταματήσω να μιλώ τώρα. Νομίζω ότι θα ελπίζω ότι θα έχω την υποστήριξη των πολιτικών ομάδων με ιδέες και προτάσεις ώστε όπως είπα να φτιάξουμε τελικά μια στέρεη και στεναρή γνωμοδότηση. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα, επομένω, όλα αυτά αποδείξατε ότι τα έχετε τεκμηριώσει, τα έχετε μελετήσει και όπως είπατε, όσο πιο νωρίς διεκπεριώσουμε την εργασία μας, τόσο το καλύτερο και τώρα οι σκιώδεις εισηγητές, αν θέλουν να λάβουν το λόγο. Κυρία Μάνερ, πρώτη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε την εισηγήτρια γιατί για άλλη μια φορά δούλεψε πάρα πολύ καλά. δεν και δύσκολο να συμφωνήσει κανείς με την εισηγήτρια. Πάρα πολύ ξεκάθαρα μας τα είπε. Και, όπως είπε, θέλουμε να διατηρήσουμε τουλάχιστον το τρέχον επίπεδο χρηματοδότησης και για το μέλλον. Επίσης, πρέπει να μπορέσουμε να ξεδιαλύνουμε κάποια άλλα θέματα τα οποία αποτελούν προτεραιότητες. Και εγώ συμμετέχω στην Επιτροπή ΣΟΥΡ και θα πρέπει να δούμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία που μπορούμε να αποκτήσουμε για την ε, στρατηγική ενώ του 2020. Άρα εδώ έχει σημασία η πολιτική συνοχή. Δεν θα βλέπουν τα πράγματα μαύρο-άσπρο. Μερικοί θεωρούν ότι η πολιτική συνοχή είναι μόνο η έκφραση αλληλεγγύης. Δεν είναι αλήθεια αυτό γιατί θα πρέπει να δούμε τη σχέση μεταξύ πολιτικής συνοχής και φυσικών πόρων, καινοτομία, ε, οικολογικής ε, συμπεριφοράς. Όλα αυτά είναι περιφερειακή πολιτική και να μην ξεχνάμε την έρευνα και ανάπτυξη. Όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Και βέβαια μπορούμε να αυξήσουμε την πρικοδότηση, αλλά να προσέξουμε να πετύχουμε τους στόχους για το 2020. Να βλέπουμε δηλαδή το ευρύτερο σκηνικό. Οι περιφέρειες στόχου 1 και 2 θα πρέπει να συνεχίσουν να χαρακτηρίζονται τέτοιες και όσον αφορά την προσθεμένη αξία θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς θα προβληθεί αυτή η προστεμένη αξία με την πολιτική συνοχή. Πώς δηλαδή ο κόσμος θα βλέπει τα προγράμματα και τα έργα που έχει χρηματοδοτήσει η Ένωση. Και αυτό είναι σημαντικό και να μην το ξεχνάμε. Επίσης, όσον αφορά την επανεθνικοποίηση της πολιτικής συνοχής που σε κάποιους κύκλους έχει αναφερθεί, αυτό θα πρέπει να το καταπολεμήσουμε είναι πολιτική πολύ σημαντική, θα πρέπει να παραμείνει πολιτική της Ένωσης. Όσο γίνεται περισσότερο. Γιατί έχει συμβάλει στο να αλλάξει η ζωή του κόσμου. Τώρα όσον αφορά το σχετικό ταμείο, το Ταμείο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, Και εκεί θα πρέπει να βρούμε ένα μοντέλο για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου και οι πολιτικές συνοχής προχωρούν παράλληλα μην υπάρχει κατάτμιση, μην αρχίσουμε να έχουμε ξεχωριστό ταμείο για τις μεταφορές, γιατί αυτό θα μπερδέψει τα πράγματα. Και θα είναι κακό και για τη χρηματοδότηση τώρα όσον αφορά την περίοδο της χρηματοδότησης. Συμφωνώ ότι πενταετία δεν αρκεί. Και από την μεριά το 5 συν 5, 10 είναι περιβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλλον τα 7 έτη είναι η πιο σωστή λύση. Αυτά για την έκθεση. Και θα κάνω την μπορώ για να συνεργαστούμε όσο είναι πιο στενό με την ε, εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Όντως πρέπει να δουλέψουμε για μια πολύ σημαντική έκθεση. Οι προθεσμίες είναι σύντομες και είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα και να εμβαθύνουμε διότι είναι μια γενική συζήτηση που αφορά το πολιετές ε, χρηματοδοτικό πλαίσιο και σήμερα καθορίζει κατά κάποιο τρόπο το μέλλον και τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, παίξει ρόλο για την ευημερία και το μέλλον των συμπολιτών μας. Πολλά ζητήματα μπορούμε να ε, θέσουμε. Εμείς θα θέλαμε να θέσουμε το θέμα της αλληλεγγύης, ότι η αλληλεγγύη δεν είναι μόνο μια κατανομή του πλούτου. Η Ευρώπη που δεν θα θέλαμε είναι μια Ευρώπη που να συγκεντρώνει όλες τις δραστηριότητες σε ορισμένες ζώνες, σε ορισμένες περιφέρειες που είναι πολύ γνωστές στον άξονα Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο, Μιλάνο και αγνοεί το υπόλοιπο την υπόλοιπη ευρωπαϊκή επικράτεια. Βλέπουμε ότι αυτή η μου συνοχή της ευρωπαϊκής επικράτειας δεν είναι και εκτιμένο. Όταν περνάμε από το Παρίσι στα βάθη της βουλγαρικής εξοχής, όπου βλέπουμε ακόμα ότι οργώνουν με τα ζώα, ε, διαπιστώνουμε ότι είμαστε στην ίδια Ήπειρο και είμαστε ε, με έναν αιώνα διαφορά. Πρέπει λοιπόν να μπορέσει και αυτή η περιοχή να αναπτυχθεί Υπάρχει μια, ένα μέλλον λοιπόν για την πολιτική συνοχή και από την άλλη πλευρά πρέπει να ε, ε, σκεφτούμε τους στόχους της. Όταν δεν υπάρχουν πια περιφέρειες κάτω από το 75 του ΑΕΠ ενώ άλλες περιφέρειες είναι στο 150% ε, του ΑΕΠ όπως η περιοχή του Παρισιού για παράδειγμα σημαίνει αυτό πως έχουμε φτάσει σε συνοχή, Ευρώπη με συνοχή ή μήπως θα πρέπει να κλείσουμε τις... Ε, ε, να, μειώσουμε ακόμα περισσότερο τις διαφορές ώστε να έχουμε ένα στάνταρ ευρωπαϊκό το οποίο να μπορεί να προσφερθεί σε όλους τους ε, Ευρωπαίους πολίτες όπου και αν κατοικούν. Και όποιος και αν είναι ο πλούτος της περιφέρειας στην οποία έχουν γεννηθεί. Και εδώ τίθεται και το θέμα των πόρων. Νομίζω πως η πολιτική συνοχή είναι αυτή που δίνει τα περισσότερα επιχειρήματα ώστε να μην πειρασπιστούμε τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η λογική που λέει ότι η Ευρώπη πρέπει να χρηματοδοτείται από ένα ποσοστό του ΑΕΠΑ ανακάτοικο στέκει αν θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να ανακατανύμουμε τους πλούτους προς τους πολίτες που είναι πιο στερημένοι μέσω της στηρίξης του εισοδήματος των γεωργών κτλ. Όμως, αν θέλουμε να επανεσορροπήσουμε την ευρωπαϊκή οικονομική δραστηριότητα, εκεί βρισκόμαστε σε ευρωπαϊκή επικουρικότητα. Σε ένα τομέα δηλαδή όπου τα κράτη, ανεξάρτητα τα μεν των δε, δεν έχουν τη δυνατότητα να μετρήσουν το πρόβλημα στα πραγματικά μεγέθη. Αυτοί οι πόροι εξάλλου ε, μπορούν να οδηγήσουν και να οθήσουν άλλες πολιτικές. Δηλαδή, αν είχε γίνει προσπάθεια στους καλούς τομεί, στους σωστούς τομείς και εμείς προτείνουμε φορολογία στον άνθρακα για παράδειγμα, ε, θα είχαμε ένα αποτέλεσμα μόνο της, ε, της εκτέλεσης του πόρου, πριν να προχωρήσουμε στην εκτέλεση της δαπάνης. Γι' αυτό και προτείνουμε να ε, δημιουργήσει η Ευρώπη ίδιους πόρους δικούς της Φόρος του άνθρακα λοιπόν, περισσότερο από ό,τι άλλα εργαλεία που προτείνει η Κομισιόν σε ένα είδος καταλόγου, αλλά νομίζω θα πρέπει να επιμείνουμε ώστε να προχωρήσουμε προς φορολογικά εργαλεία που τα ίδια ε, θα βοηθήσουν στην επιτυχία στο μέλλον. Αυτά Πρόεδρε. Εμείς ε, περιμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια αυτής της εργασίας και φυσικά θα είμαστε παρόντες. Να, συγγνώμη, ε, ξέχασα να ε, το πω. Θέλουμε να επιμείνουμε και για τον σημαντικό χαρακτήρα των διαμεθοριακών συνεργασιών, γιατί και νομίζω πως και εκεί έχουμε ένα πολύ σημαντικό κοίτασμα ανάπτυξης για την Ευρώπη και τους πολίτες της. Και συχνά με σε αυτή την κληρονομιά της περίοδου πριν την Ευρώπη, όταν δηλαδή τα σύνορα ήταν φέοδο κάθε κρατικής μόνο δαπάνης, βλέπουμε και ακριβώς και τη σπατάλη, τη σπατάλη. Τα νοσοκομεία δεν τα μοιράζονται από τις δύο πλευρές των συνόρων, τα δύο μεγάλα αεροδρόμια από τη μια πλευρά των συνόρων και από την άλλη, ε, ακριβώς επειδή το κάθε κράτος έκανε του κεφαλιού του. πρέπει λοιπόν να υπάρξει κοινοτική ε, πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σον Κέλλη. Καταρχήν, θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια που έκανε μια εξαίρετη σύνοψη για το πού βρισκόμαστε και ίσως το πού πρέπει να προχωρήσουμε, προς πού πρέπει να οδεύσουμε. Είναι δύσκολα θέματα αυτά. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε επί της ουσίας και γρήγορα. Κάποιες παρατηρήσεις που έκανε απήχησαν τα όσα ακούσαμε σήμερα το πρωί από την κυρία Σάντσε Σμιτ στην εξέταση της έκθεσής της. Καταρχήν μίλησε για διαφορά στις δαπάνες, ανισότητα στις δαπάνες, στην χρηματοδότηση συνοχής, 250 εκατομμύρια ευρώ στο στόχο 1, 49 δις για το στόχο 2 και μόνο 7,5 για τον στόχο 3 που είναι 2,5%. Από την άποψη της ε, συνεργασίας ε, των ε, περιφερειών και την ανάπτυξη της θέσης ότι η Ευρώπη υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί οι αριθμοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και ίσως να πρέπει να γίνουν και κάποιες προσαρμογές καθώς προχωρούμε. Ιδιαίτερα η παρατήρηση που έκανε πάλι η συγγήτρια και η κυρία Σάντζε Σμιθ για την απόλυτη έλλειψη ορατότητας από τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τα ωφέλη των όσων συμβαίνουν στην Ευρώπη με τα κοινοτικά χρήματα είναι εντυπωσιακή. Είναι εντυπωσιακό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν χρηματοδότηση ευρωπαϊκή με κάποιο τρόπο ή που οφείλουν τη δουλειά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το ξέρουν καν. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι κάνουμε εκεί, γιατί υπάρχει πολύ αρνητική ε, στάση Ούτως ή άλλως πάντοτε τα κακά νέα είναι τα καλά νέα. Δηλαδή αυτά διαδίδονται πάντα πιο γρήγορα. Ωστόσο, χαίρομαι και πάλι που γίνεται αυτή η συζήτηση. Πιθανότατα το Συμβούλιο θα έχει εδώ αντιρρήσει. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να εξετάσουμε το το θέμα εις βάθος για να δούμε και ποιες δυνατότητες θα έχουμε για να αξιοποιηθούν όλα αυτά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή συζήτηση αλλά και διαφήμιση. Διαφήμιση ώστε να περάσουν αυτές οι ιδέες. Τέλος. Τώρα αν είναι πενταετία, εφταετία, δεκαετία, εφτά νομίζω εγώ λιγότερο. Και είμαι πεπισμένος ότι τα δέκα χρόνια θα ήταν το καλύτερο. Αυτά ευχαριστώ. Σρέτερ. Πρώτα ευχαριστώ και εγώ την Κωνσταντσε για την ε, πρώτη αυτή ε, εισήγηση. Πράγματι χρειάζεται πολλή δουλειά. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά που θα πρέπει να αγωνιστούμε υπέρ των θέσεών μας και απέναντι στην Επιτροπή ΣΟΥΡ και απέναντι στην Επιτροπή Προπολογισμών. Για τις προτεραιότητες, για παράδειγμα, για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, για το θέμα επίσης που θα πρέπει να μπουν τα όρια των χρηματοδοτήσεων Και εκτός από τα θέματα αυτά, βέβαια, να σκεφτούμε και το, αν θα βάλουμε δηλαδή και το θέμα της εφαρμογής. Ακούσαμε ότι θα υπάρξει κοινή ρύθμιση των ελέγχων. Μήπως λοιπόν πρέπει να μπει και αυτό το θέμα εδώ για να αξιολογηθεί. Αλλιώς δεν βλέπω πού μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα εκ των προτέρων να θέσουμε τα θέματα αυτά εάν όχι μέσα στα πλαίσια ένας τέτοιου ψηφίσματος. Και το άλλο ερώτημα που τίθεται είναι τι γίνεται όταν δεν απορροφώνται τα κονδύλια ή εάν καταλήξουν εν τέλει σε κάποιο άλλο τμήμα του προπολογισμού. Τι θα πρέπει τότε να κάνουμε. Αυτά βέβαια δεν μπορούμε τώρα να τα συζητήσουμε επί της ουσίας, αλλά είναι θέματα τα οποία έχουν ε, μεγάλη σημασία και εμείς είμαστε υπέρ της συγκέντρωσης, αλλά να μην δίνονται χρήματα τα οποία να παρεμποδίζουν άλλες κοινοτικέ πολιτικές. Αυτό για μας τους πράσινους είναι πολύ σημαντικό. Άλλος κανείς? Εσείς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να προσθέσω δύο λόγια. Γιατί ήταν πλήρης η εισήγηση της κυρίας Κλέρ να δούμε τι γίνεται όσον αφορά αυτήν την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της συνέχειας. Για να υπάρχει συνέχεια, πιστεύω ότι χρειάζεται η κατάλληλη χρηματοδότηση. Να έχει καθοριστεί για το μέλλον ξεκάθαρα αυτή. Να τεγνήσουμε μένω στο μέλλον, να το συζητήσουμε και να καθορίσουμε πώς θα βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των επιμέρους στόχων που έχουμε τάξει για το μέλλον. Δηλαδή, αηφόρος ανάπτυξη για τις πόλεις, αλλά και για την Ήπεθρο. Θα πρέπει η πολιτική συνοχή να συνεχίζει να καλύπτει την Ήπεθρο. Γι' αυτό θέλω να σας αναφέρω και τα έργα υποδομής, να καταβληθεί επομένως προσπάθεια όσον τα έργα υποδομής. Φυσικά και θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης. Συμφωνώ για το ότι θα πρέπει να έχουμε αυτήν την επταετία και για, μετά το 2013 θα πρέπει να εντάξουμε την υπόθεσή μας στα πλαίσια της πολιτικής της Ευρώπης για το 2020. Ευχαριστώ λέει η πρόεδρος θέλει κάποιο άλλο το λόγο γιατί έχουμε ακόμη ένα-δύο θεματάκια από ό,τι έχω καταλάβει. Σε αυτή την έκθεση δεν πρέπει να ασχοληθούμε με το όλο όραμα του μέλλοντος για αυτή την πολιτική. Θα πρέπει να εντάξουμε την πολιτική αυτή στα πλαίσια του προϋπολογισμού για το μέλλον. Όχι μόνο από πλευράς ε, ταμείων, πόρων, αλλά ως συνόλου πολιτικών που θα πρέπει να αποδώσουν κάτι όσον αφορά τους στόχους της Ευρώπης και για αυτό θα πρέπει να είμαστε αρκετά αποφασιστικοί για να αναδειχθεί αυτή η προστιθέμενη αξία. και με τις πολιτικές αυτές να έχουμε και τον κατάλληλο μηχανισμό ούτως ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος και σταθερός μηχανισμός για κάθε επίπεδο διακυβέρνησης και για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε όσα πραγματικά χρειάζεται η Ευρώπη για να γίνει η ζωή των Ευρωπαίων καλύτερη στο μέλλον. Να αντιμετωπίσουμε τις αντίστοιχες προκλήσεις και είναι σημαντικό αυτό το οποίο ελέγχθη από πολλούς συναδέλφους ότι θα πρέπει να τοποθετηθούμε όσον αφορά το timing για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, για τις επόμενες χρήσεις της μεσονομικές. Η Επιτροπή μας βεβαίως και στοχεύει καταρχήν στην πολιτική συνοχή, η οποία όμως για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να ενταχθεί στον προπολογισμό, όχι μόνο από πλευράς πρικοδότησης, <clears throat> αλλά και από πλευρά διάρθρωσης του προπολογισμού. Αν λοιπόν η διάρθρωση είναι αν υπάρχει μια κατάτιμηση στον προπολογισμού για το τι κάνει ο καθένας, αυτό δεν μα εξυπηρετεί με έναν τέτοιο εξειδικευμένο το συμπίνη προπολογισμό. Θα πρέπει οι στόχοι ε, το 2020 να αντιστοιχούν και να αντικατοπτρίζονται στον προϋπολογισμό. Αυτά ως γενικές παρατηρήσεις. Και από την πρόκληση επίσης, αυτό που συζητάει, τρεις προηγούμενες με κάποιους αδέλφους, το τι συζητείται όσον αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές. 5 το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν 5 συν 5. Το 7 μάλλον δεν ισχύει πια. Αν και βέβαια η πολιτική μας εξυπηρετείται από την επταετή περίοδο. Άρα ίσως θα πρέπει να επανέλθει στο τραπέζι των συζητήσεων. Και να δούμε τι θα πετύχουμε. Και βέβαια το εναλλακτικό σενάριο να είναι το 5 συν 5. Αλλά το 5 συν 5 απλώς διπλασιάζει τα προβλήματα του 5 δεν είναι λύση επομένω. Άρα θα πρέπει στα σοβαρά να καταπιαστούμε και με αυτό. Επίσης θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους τους συναδέλφους με είναι τόσο σημαντική αυτή η έκθεση. Όχι μόνο να βοηθήσουμε τον, την εισηγήτρια, αλλά να υπάρξει συνεργασία όλων των πολιτικών ομάδων. Να μην έχουμε αγκάθια ιδεολογικά. Να μην είναι λοιπόν μια έκθεση της κυρίας Κρέλ αυτή, να είναι έκθεση της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Πολιτικής. Συμφωνώ και εγώ και σας συγχαίρω κυρία Συγγετρία. Σήμερα δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο χρονοδιάγραμμα, δεν ξέρουμε ακόμα το πλαίσιο, αλλά πρέπει να ψηφιστεί σχετικά άμεσα. Δεν έχουν πολλά χρονικά περιθώρια επομένω. Όλμπριχτ. Δεν έλαβα το λόγο και δεν άκουσα όλη την εισήγηση, αλλά η πολιτική απόφαση είναι το τι θέλουμε. Να έχουμε τελειώσει πριν καταλήξει η Επιτροπή Σούρε ή μετά. Γιατί έχουμε την Σούρε που θα ασχοληθεί με αλληλεγγύη και συνοχή. Για να προσέξουμε καλύτερα ή ίσως να ξέρουμε περισσότερα από την μέσα Διάταξη στην επόμενη μας συνεδρία. Τι θέλουμε, θέλουμε να αντιδράσουμε σε ηλυμένη απόφαση, θέλουμε να την προκαταλάβουμε. Ε, Σρέντερ, συγγνώμη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Γιάνν. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει εδώ όσο γίνεται περισσότερο να το συζητήσουμε, αλλά να τηρήσουμε στάση αναμονής για το τι θα γίνει στην Σούρα. και να προσαρμόσουμε τις τροπολογίες μας αναλόγως. Αφού καταλήγουμε στα βασικά σημεία και συμφωνήσουμε και πριν ψηφίσουμε να γίνει ζήτηση στη Σούρα και ενδεχομένω να έχουμε φυσικέ αντίστοιχε ανάλογε τροπολογίες ή συμβαστικέ τροπολογίες. Και μετά να πάμε για την ψήφιση της δική μα έκθεση. Δεν ξέρω, Κωνσταντ, τι έχει να πει. Κωνσταντ. Η κυρία Κρέλ. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται όντως μια εντατική συζήτηση στην Επιτροπή μας εδώ, που νομίζω ότι μπορεί να διεξαχθεί τον Δεκέμβρη και με την θέση που θα προκύψει από την συζήτηση αυτή, που θα την βάλουμε και στο σχέδιο γνωμοδοτήσεως και θα υποβάλουμε μετά στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ, να δούμε όμως και από αυτούς τι θα προκύψει. Έχω την εντύπωση ότι εδώ στην Ευρωβουλή ο καθένας γνωρίζει, επειδή όλοι προέρχονται από κάποια περιφέρεια, γνωρίζει τι λεπτομέρειε τουλάχιστον ενό έργου στην περιφέρειά του. Αυτό είναι σωστό και καλό. Αλλά όλες αυτές τι προφορίες μαζί οδηγούν κάπως σε σύγχυση. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε προσεκτικά. Υπάρχει ίσως μια ιδέα που αρχίζει και διαμορφώνεται από τι εργασίε τη επιτροπή ΣΟΥΡΕ και στην οποία ιδέα θα πρέπει κανεί να βγει και να απαντήσει, να πούμε γίνεται ή δεν γίνεται, ξέρω εγώ. Αυτό με τα 100% χρηματοδότηση, για παράδειγμα, που άκουσα σήμερα και μου προκάλεσε πραγματικά ε, μια σχετική σύγχυση. Ε, όπως είπα, θα υποβάλω και τροπολογίες. Και στον χρόνο που διαθέτουμε μέχρι τότε, ε, θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε και σε ορισμένα πράγματα που παράγει η Επιτροπή ΣΟΥΡΕ. Η πρόεδρος Χιούπνερ. Πάντα είναι καλύτερα να επηρεάζει κανείς εκ των προτέρων παρά να αντιδρά εκ των υστέρων. Γιατί η εμπειρία που με διδάσκει από τη δραστηριότητά μου και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι όταν κάτι έχει πλέον τεθεί είναι δύσκολο να ε, τροποποιηθεί. Βέβαια, εμείς επηρεάζουμε και ε, την, ε, τις απόψεις του εισηγητού της Επιτροπής ΣΟΥΡ λαμβάνοντας τον λόγο στην ίδια την Επιτροπή ΣΟΥΡ και διατυπώνοντας ε, τις προτάσεις μας. Θα διαβιβάσω στην ε, πρόεδρο της ΣΟΥΡ, Γιούτα Χάουκ, όλα τα έγγραφα που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα και θα δούμε όταν θα υποβάλει το σχέδιό της η Κωνσταντσε Κρέλ θα δούμε μετά με ποια ταχύτητα μπορούμε να προχωρήσουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι. Και επίσης σύμφωνα και με τα όσα λέει η ε, κυρία Σρέντερ, θα έχουμε τη δυνατότητα ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, να ζητήσουμε από την Επιτροπή Σούρε να αντιδράσει και να διαμορφώσει και το χρονοδιάγραμμά της, σύμφωνα λίγο και με το δικό μας. Αν δεν επιθυμείτε να, να πείτε τίποτε άλλο, Κωνσταντσε, τότε νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο... Α, παρακαλώ, με συγχωρείτε, Γιάννη μια σύντομη πληροφορία που είναι χρήσιμη για την Επιτροπή μας, να συμμετάσχει δηλαδή στην ακρόαση που θα γίνει στην Επιτροπή ΣΟΥΡ, όπου το 1 τρίτο της ακρόασης αυτής θα είναι σχετικά με τη συνοχή και νομίζω είναι στις 28 Νοεμβρίου. Ορισμένοι από τους εμπειρογνώμονες θα είναι ε, ο Μπάρκα και ο Σαπίρ στα διάφορα πάνελ. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και για τη δική μας Επιτροπή να με, να ακούσουμε τις απόψεις τους. Η κυρία Χίπνερ, όπως με έχουν πει και οι συνάδελφοι μας της Κομισιόν, υπάρχει μια καλή πρόταση από την Κομισιόν, πρέπει να την παρακολουθήσουμε, να συνεχίσουμε να διατυπώνουμε τις απόψεις μας και για το μέλλον, διότι όντως λαμβάνονται υπόψη και από άλλα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ, θα σας δώσω τις τρεις.